Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα θυμάστε ότι περίπου πριν από ένα χρόνο είχαμε μία συνάντηση με νέους και τότε συζητήσαμε την εκλογική νομοθεσία. Και μας ζήτησαν να μειώσουμε την ηλικία ε, εκλογής στα 16 χρόνια, ειδικά στον Αυστριακό συνάδελφο. Αναλάβαμε αυτή τη δέσμευση και το συμπεριλάβαμε στο προσχέδιο κειμένου, όμως απορρίφθηκε η ιδέα αυτή να μειωθεί το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Εμείς Το έχουμε στην Αυστρία σαν πρόταση και αλλού ίσως στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο εν ώψη του δημοψηφίσματος υπήρχε αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, φέτος, σήμερα δίνουμε συνέχεια με, στην συνεδρίαση που έγινε ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεότητα, η οποία έλαβε χώρα στο Στρασβούργο 20 και 21 Μαΐου, όπου συζητήθηκε η πολιτική στην Ευρώπη, η δημοκρατία και άλλα θέματα καταρχάς και όλο τον Οκτώβριο και όλο τον Νοέμβριο έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακροάσεις και συναντήσεις με τους ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει στο φόρουμ του Στρασβούργου του Μαΐου. Αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να ακούσουμε τις ιδέες τους για διάφορα ζητήματα και διάφορες απόψεις που είναι πολύ σημαντικές και για εμάς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εν συντομία να σας συστήσω τους τρεις συναδέλφους. Πρώτον, εξ αριστερών μου, ο κύριος Νικολάους Έρλιγκερ, δευτεροετής Φοιτητή από την Αυστρία. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε μπορείτε να πάρετε το λόγο. Είστε φοιτητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Έχουμε τη Λεόνι Σλότς, στη συνέχεια από τις κάτω χώρες, πρώην φοιτήτρια. Δεν είστε πια φοιτήτρια, είστε από τις κάτω χώρες και ζείτε στο Ενωμένο Βασίλειο. Και εργάζεστε στο Ενωμένο Βασίλειο. Και όχι μόνο είστε πτυχιούχος νομικής, αλλά είστε και συνθέτης και τραγουδίστρια. Καλό είναι να έχει κανείς και άλλες επαγγελματικές διεξόδους, εάν χάσει τη θέση εργασίας του. Μπορείτε και να μας τραγουδήσετε. Έχουμε και την Σέγια Ακίουαβο από το Ηνωμένο Βασίλειο, που εργάζεται σε ένα από τα Δημοτικά Συμβούλια του Λονδίνου. ουσιαστικά ανήκεται στη Βρετανική τοπική αυτοδιοίκηση, εξ όσων γνωρίζω. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι έχουμε δύο συναδέλφου με ισχυρού δεσμού με το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, γιατί έτσι μπορούμε να μάθουμε περισσότερα και αυτό ε, θα δώσει μια έντονη νότα στις συζητήσεις μας. Βασική ιδέα είναι να έχουμε ερωτήσεις από τους συναδέλφους και αντιδράσεις και απαντήσεις από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω σε τρεις θεματικούς άξονες. Πρώτον, το μέλλον της Ευρώπης μετά το Brexit. Δεύτερον, ενεργή δράση του πολίτη. Και τρίτον, συμμετοχή των νέων πιο ενεργητική στην Ευρώπη του, και αξιοποίηση του προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Νεολαία. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός, πρέπει να είμαστε επιθαρχημένοι στην έκφρασή μας Παραδοσιακά το Κοινοβούλιο δίνει 2-2,5 λεπτά στον καθένα, κατ' εξαίρεση μπορεί κάποιος να πάρει 5 λεπτά και στην Ολομέλεια βεβαίως λιγότερα ενδεχομένω, για να μιλήσουν και περισσότεροι. Έχουμε τη συνήθεια λοιπόν να είμαστε επιθαρχημένοι. Στρέφομαι προς τους προσκεκλημένους και τους ζητώ να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους για αυτά τα τρία ζητήματα ο ένας μετά τον άλλον, οι τρεις ομιλητές και στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής μας, βουλευτές, θα ε, σχολιάσουν αυτές τις ιδέες. Ξεκινούμε με τον πρώτο άξονα, το θεματικό, το μέλλον της Ευρώπης μετά από το Brexit. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες στην Ευρώπη και όχι μόνο στις Βρυξέλλες. Όλοι συζητούν για το τι συμβαίνει τι μπορεί να συμβεί εάν ε, προκύψει το Brexit. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νέοι αρνήθηκαν να πούν ναι να φύγουμε. Ε, με μεγάλη πλειοψηφία η δική σας γενιά 18-24 ψήφισε υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεωνί Σλότς, θα είστε η πρώτη. Έχετε δύο λεπτά να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι το σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης μετά το Brexit. Θέλω να μιλήσω για το δικαίωμα πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διαδικασία στην δεν αρκεί. Εάν θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτε να ξανανακτήσουν την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Brexit ε, επώδυνα απέδειξε ότι η πλειοψηφία των Βρετανών δεν πιστεύουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αρνούμαστε την αλήθεια αν πιστεύαμε ότι αυτό αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξανασκεφτεί τι μεθόδου τη, δεδομένου του δικαιώματος πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήταν ένα πρώτο βήμα αυτό για να εκπροσωπήσουμε πραγματικά τη θέληση των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπλέκεται συχνά σε πολύ τεχνικά θέματα και είναι πολύ μακριά από τους Ευρωπαίους πολίτες για να γνωρίζει τι χρειάζονται. Παρότι οι πρωτοβουλίες αυτές συζητώνται με όλους τους φορείς, πριν οδηγήσουν σε πραγματική πρόταση, δεν αρκεί αυτό για να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι ευρωπαϊκές φωνές ακούγονται. Με το δικαίωμα πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να αντιδράσει σε πολλά θέματα. Από τη μία θα μπορεί άμεσα να εξετάζει θέματα εκλογικών περιφερειών και να αυξηθεί το αίσθημα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι ακούγονται και ότι μετράνε. Από την άλλη θα αυξηθεί η διαφάνεια και η νομιμότητα Τη Ευρωπαϊκή Νομοθετική Διαδικασία. Η πρωτοβουλία για την νομοθεσία θα είναι η βασική ευθύνη των εκλεγμένων εκπροσώπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και των Ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα. Ένα άλλο πλεονέκτημα ε, θα βελτιώσει τον πραγματικό πολιτικό διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προτάσει νόμου. Αυτό θα αυξήσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της ε, διαδικασία της νομοθετικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ πιστεύω ότι το δικαίωμα πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας εξασφαλίσει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο μιλητή. do it often, so you Δεν χειροκροτούμε συχνά, μάλλον το αξίζεται αυτό το χειροκρότημα. Πάμε τώρα στον Νικολά για να μας πει και αυτό στις ιδέες του. Η πρότασή μου είναι να ανοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να έχουμε μια αλλαγή προς μια πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαφάνεια. Αυτό αφορά δύο θέματα. Το πρώτο είναι η εφαρμογή μιας υποχρεωτικής καταγραφής των λόμπις και ένα ε, βιβλίο επισκεπτών των ε, θεσμικών όργανων. Αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλοί σήμερα θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνεια και δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την λήψη αποφάσεων. Οι αποφάσει δεν εκπροσωπούν πάντα τη βούληση των ε, πολιτών. Και γι' αυτό πολλοί φοβούνται ότι αυτοί που έχουν ισχύ μπορούν να προωθήσουν νομοθεσία από την πίσω πόρτα. Και αυτό δημιουργεί μια τέτοιου είδου ατμόσφαιρα στο κοινό και προωθεί και δίνει έδαφο ε, στην πραγματοποίηση ακραίων σενάριων όπω είναι το Brexit. Η υποχρεωτική καταγραφή των λόμπι, ένα α, ε, μητρό διαφάνεια θα βοηθήσουν να υπάρξει διαφάνεια στην νομοθετική διαδικασία. Επίση, συνεδριάσει των ε, συμμετεχόντων σε λόμπι με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μπορούν ε, να ε, καταγράφονται και να ακολουθούνται μέσα από ένα σύστημα. Ένα δεύτερο θέμα είναι να υπάρξουν διαβουλεύσεις με τους πολίτες σε μια online πλατφόρμα και σε, ανοιχτά, σε εκδηλώσεις για να θυχτούν αυτά τα θέματα στο κοινό που αφορούν το, μέλος, ε, το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση οι πολίτες με την εφαρμογή και τη δημιουργία διαβουλεύσεων μέσω online ε, πλατφορμών ε, και μέσω εκδηλώσεων που θα μπορούν να λάβουν χώρα τέτοιου γεγονότα, π.χ. είτε στο Ευρωκοινοβούλιο και θα είναι ανοιχτά στο κοινό ώστε να μπορούν να συζητήσουν την ε, διαδικασία τη νομοθεσία. Θα είναι έτσι μέρο τη διαδικασία και οι πολίτε και θα μπορούν να μοιραστούν τι απόψει του για διάφορα θέματα και έτσι να επαναγκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Νικολάου. Και δύο ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την ε, εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Νομίζω ότι είστε, κινείστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτά τα θέματα τα οποία θέξατε δεν ε, μα απασχολούν πάρα πολύ και δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ασχοληθούμε με αυτό το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να πάρει το λόγο ο κύριο Κόρμπετ, Μα παρουσιάστηκαν δύο ιδέε τώρα, μπορούμε να δώσουμε την απάντησή μα τώρα και μετά να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Ο λόγο των Τζόρτζ. Μια πρώτη αντίδραση. Και σου θυμίζω ότι έχει δύο λεπτά, λέει Πρόεδρο. Υπάρχει περιορισμό ε, στον χρόνο για να έχουμε τι ευκαιρίε εδώ. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση πολύ στον επιχείρημα όσον αφορά την ε, πρωτοβουλία όταν γίνονται εκλογές για το Κοινοβούλιο περιμένουμε να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους. Υπάρχουν προσδοκίες. Όσον αφορά το δικαίωμα πρωτοβουλίας Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ασκήσουμε πίεση στην Επιτροπή αν δεν προωθήσει κάποια θέματα. Δεν θα ήταν άσχημα να το συγκρίνουμε αυτό με κάποια εθνικά κοινοβούλια όπως είναι το δικό μου, όπου υπάρχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και υπάρχει ένα σύστημα για κάποια νομοσχέδια τα οποία πολλές φορές δεν υιοθετούνται. Έχετε δίκιο όπως και να έχει, όμως πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα όσον αφορά τη διαφάνεια. Συζητήσαμε γι' αυτό σήμερα το πρωί. Μιλήσαμε για τον εσωτερικό κανονισμό ε, που θα πρέπει να ευθυνθεί τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει ένα πακέτο μέτρων που αφορούν ε, την διαφάνεια. όσον αφορά ε, την ομφυλική διαδικασία να καταγράφουν τα άτομα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή οι ευρωβουλευτές για το ποιος μπορεί να εισέλθει στους χώρους του Κοινοβουλίου κτλ. Αν δείτε όλα αυτά τα νέα ε, στοιχεία που έχουμε για τον ιστορικό κανονισμό, θα είστε αρκετά ευχαριστημένους και πιστεύω ότι έχει γίνει πρόοδο σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. George, you wanted. Και ο George θα θέλει να πάρει το λόγο. Δεν ε, το είπα, συγγνώμη. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ ανήκει στην ομάδα των σοσιαλιστών και ο Τζορτ Σέπλιτ είναι και Ούγγρος και Βρετανός. Είναι από το ΕΛΚ. Καλώς ορίσατε. Έχω διάφορες σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Καταρχάς, σε σχέση με το δικαίωμα ίδιας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως το ανέφερε η Λέωνη Σλότς. Πιστεύετε ότι υπάρχει και ότι θα έπρεπε να υπάρχει ε, ένα ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής και αν ναι, πώς αυτό αλληλεπιδρά με το εθνικό επίπεδο πολιτικής. Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα. Και όταν γίνεται λόγος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κόσμου στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σας ρωτώ, υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα, διότι αν δεν υπάρχει, τότε είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν θα πάμε και πολύ μακριά. Προς τον κύριο Έντλιγκερ τρέφομαι τώρα για να πω το εξής. Η βούληση του λαού ε, την οποία αναφέρεται είναι και ο λόγος που συχνά έχετε κανείς κατηγορίες για λαϊκισμό. Ε, γίνεται μια πολύ σοβαρή συζήτηση αυτή τη στιγμή και Πολύ συχνά λέγεται ότι όποιος μιλάει για τη βούληση του λαού ε, και για την ύπαρξη του λαού, τότε συνεχώς τον αποκαλούν λαϊκιστή. Δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά οφείλετε να το έχετε υπόψη σας. Από εκεί και πέρα, η εμπιστοσύνη... Ε, ε, ε, σχετίζεται πολύ και με την έλλειψη εμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν κανείς αποκαλύπτει κάτι, δημιουργεί το εξή ερώτημα. Πόσα πολλά είναι κρυμμένα από πίσω που δεν μάθαμε ακόμα. Θα έλεγα το εξή. Έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι να είναι πολιτικώς ουδέτεροι. Θα έπρεπε να έχουν πολιτικό κίνητρο και με αυτά ολοκληρώνω γιατί έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Έχουμε την επόμενη συνάδελφο από τους σοσιαλιστές Ιταλίδα. Θα μιλήσω Ιταλικά, γι' αυτό σας παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Εάν δεν μιλάτε Ιταλικά βεβαίως. Ε, ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και από πλευράς μου για τις δύο παρουσιάσεις που ακούσαμε. Για την πρώτη παρουσίαση, το δικαίωμα πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα σημαντικός περιορισμός που τον αισθανόμαστε και εμείς στο πετσί μα. Και στις δύο εκθέσεις που ετοιμάζει η δική μας Επιτροπή, επευκαιρία των, της εξικονταετίας από τη συνθήκη της Ρώμης που θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, μέσα στην έκθεση Φερχόφστατ, που είναι μία από τις δύο εκθέσεις, μιλάμε για τις πιθανές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στις συνθήκες. Εκεί ακριβώς αναφέρεται το, το δικαίωμα πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κάτι άλλο που είναι περίπλοκο και είναι υποσυζήτηση, τη δυνατότητα να υπάρχει μία πράσινη κάρτα ενδεχομένως για τα εθνικά κοινοβούλια, για να προτείνουν όχι κείμενα, αλλά ιδέε, όχι νομοσχέδια ή νόμους, αλλά ιδέε. Να, δηλαδή, να, να δώσουμε δηλαδή ένα δικαίωμα πολιτικής πρωτοβουλία στα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι πιο αμφισβητούμενο θέμα, αλλά ενδιαφέρον. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα. Για να προσθέσω κάτι τώρα για την διαφάνεια, που είναι ένα θέμα επί του οποίου εγκύπτει πολύ το Κοινοβούλιο. Υπάρχει μία έκθεση που είναι υποσυζήτηση, με όλα αυτά που ακούσατε από τον Ρίτσαρντ, η Επιτροπή πρόσφατα πρότεινε μια διαθεσμική συμφωνία για ένα μητρό, κοινό μητρό διαφάνειας για την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβουλίο, ένα κοινό μητρό δηλαδή. Ξεκινάμε αυτή τη στιγμή τις διαπραγματεύσεις για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Θα είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρξει μια ενιαία συμφωνία, γιατί όταν υπάρχει μια ενιαία συμφωνία είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο διαφανής, γιατί είναι αυτή, δεν χρειάζεται να ψάχνει κανείς εδώ και εκεί και, παραλού, και αλλού. Ευχαριστώ. Τώρα η Λεωνή και ο Νικολάου θα, πάρει, θα πάρουν το λόγο. Αποφασίστε ποιο θέλει να μιλήσει πρώτος. Έχετε ένα λεπτό. Η Λεωνή. Δύσκολο να σας απαντήσω στο ένα λεπτό που μου έχει δοθεί. Νομίζω όμως ότι θα προσπαθήσω να απαντήσω στα σχόλια των δύο κυρίων, διότι εσείς ε, ε, κύριε Κόρπετ και κύριε Σάλεν, μιλήσατε για τη σαφήνεια και αυτό είναι σημαντικό. Πράγματι, πολλοί δεν κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα και πολιτική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θεωρώ εκνευριστικό το γεγονός ότι μόνο Ολλανδούς μπορώ να ψηφίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι άλλους. Ε, ε, είναι δύσκολο να επιτευχθεί, είναι όμως ένα βήμα που πρέπει να γίνει. Να γνωρίσουμε και να μάθουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, να μην χρειάζεται κανείς να έχει πτυχίο στο Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό δίκαιο και ε, να μην χρειάζεται να έχει πολύ πλούσιο μορφωτικό επίπεδο για να καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το σύστημα. Ελπίζω ότι έτσι θα μειωθεί ο λαϊκισμός και θα αυξηθεί η, πολιτική, ε, η συμμετοχή στα κοινά στην πολιτική από πλευρά των πολλών. Ευχαριστώ ο Νίκολας. Ε, ευχαριστώ κι εγώ. Είπατε ότι σε σχέση με τελευταία σας δήλωση μάλλον ε, για το νομοσχέδιο και τον τρόπο με τον οποίο περνιέται, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Οι νέοι, ξέρετε, πολύ συχνά έχουν την αίσθηση ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην, ε, στα κοινά, στην πολιτική διαδικασία. Πολλοί πιστεύουν ότι η νομοθεσία τελικά μπαίνει από την πίσω πόρτα. Επομένως, δεν συμφωνώ με την ιδέα ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της εμπιστοσύνη και της διαφάνειας. Πιστεύω ότι υπάρχει. Δεν λέω ότι το ένα εξαρτάται από το άλλο. Ωστόσο, ωστόσο σήμερα αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι έλλειψη εμπιστοσύνης διότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας ή διότι υπάρχει άποψη ότι επικρατεί έλλειψη διαφάνειας. Μπορεί αυτό να οφείλεται σε εσφαλμένη επικοινωνία, δεν το γνωρίζω. Όμως ένα φαινόμενο σαφέστατο το οποίο παρατηρούμε στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, για να είμαι ειλικρινής, και η κοινή γνώμη πιστεύει ότι όλα αυτά σχετίζονται με την πολιτική. Ότι γίνονται πράγματα δηλαδή πίσω από κλειστέ πόρτε, τα οποία δεν μπορούν να ε, επηρεάσουν. Οι πολίτε δεν μπορούν να τα επηρεάσουν την έκβασή του. Νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ ενός λαϊκιστή και ενός αληθινού πολιτικού είναι ότι ο δεύτερος προσπαθεί πραγματικά να λύσει και το πρόβλημα και ελπίζω αυτό να κάνουμε. Πολύ ηχηρό το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Προχωρούμε στο δεύτερο θέμα μας. Ενεργή δράση του πολίτη όχι απαραίτητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά εσείς θα διαλέξετε ε, πώς θα το θίξετε, αν θα επικεντρωθείτε κυρίως στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες ή τις δραστηριότητες σε τοπική κλίμακα. Είναι μια πρόκληση πάντως παντού στην Ευρώπη. Έχουμε τη Σέγη Άκη Βόβο. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να μπορούμε να αποδείξουμε δείξουμε ότι η Ευρώπη ε, μπορεί να οριμάσει και να δείξει πολύ μεγαλύτερη οριμότητα από την πραγματική της ηλικία. Πολύ συχνά οι νέοι απομακρύνονται από αυτήν και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε αποδείξεις. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάξετε μια διαδικτυακή πλατφόρμα έτσι ώστε οι, νέα, νέοι Ευρωπαίοι να σας δώσουν συμβουλές και να μπορούν και να συμβουλευτούν αυτή την πλατφόρμα για τις βασικές λειτουργίες και δράσεις που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πολυμορφία και πρέπει να τη σεβαστούμε, αλλά να αναγνωρίσουμε και τους νέους από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες ή ε, από ευπα τις ομάδες του πληθυσμού, να αναγνωρίσουμε την τεράστια προσπάθειά τους προτείνω ένα διαδικτυακό σύστημα σήμερα που θα επιτρέψει ε, στους νέους, για παράδειγμα, επιθεωρητές ε, στη σχολική εκπαίδευση, επιθεωρητές σε επίπεδο ε, επιτήρησης υγείας και ασφα... και ασφάλειας των τροφίμων. Δηλαδή, να υπάρχουν συμβουλές, να, υπάρχουν, να υπάρχει ένα feedback, μια τροφοδότηση για όλα αυτά τα θέματα στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Μπορούμε να έχουμε επιτροπές, διαδικασίες, διορισμούς, και σε όλα αυτά να εμπλέκονται οι νέοι μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και κυρίως νέοι από πιο ε, δυσχερή ε, δυσχερές κοινωνικό υπόβαθρο ακριβώς για να νιώσουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την ε, δράση της θετικής διάκρισης και αν αναλάβουμε αυτή τη δέσμευση έναντι των νέων σήμερα, σε 10 χρόνια θα είναι τρομακτικά μεγαλύτερη η συμμετοχή τους στα κοινά. Θα έχουμε πολιτικές που θα συμπεριλαμβάνουν πολύ περισσότερους και θα έχουμε βελτίωση όλων των πολιτικών αλλά και των υπηρεσιών και των λειτουργιών. Ευχαριστώ. Κανάκλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εισαγάγει ένα σύστημα Ένα σύστημα λοιπόν ενεργούς ηθαγένειας ε, και την αγωγή του πολίτη στα γυμνάσια και ηλίκια, ούτω ώστε να υπάρξει ποιοτική ε, εκπαίδευση ε, στα κράτη-μέλη μέσω κατευθυντηρίων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε να δίνουμε κίνητρα στους ανθρώπους για να γίνουν πολιτικά ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτης από πολλοί νέοι. Το Brexit, ξανά πρέπει να το πω, ε, όχι μόνο επώδυνα απέδειξε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έδειξε και το μέγεθος της ε, έλλειψης κατανόησης. Ως ε, με, που ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, με πτυχίο στο, ε, στο δίκαιο, διαρωτώ με, με τι θα μοιάζει η ζωή μου όταν βγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι που ψήφισαν για τον Brexit ψήφισαν για να καταδικάσουν πράγματα που δεν είναι καν τμήμα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Για να υπάρξει μεγαλύτερη έτσι, εμπλοκή στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα ενεργού ε, ηθαγένεια, ε, εκπαίδευση των πολιτών. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ε, οι φοιτητέ, α πούμε, οι μαθητέ, πώ του επηρεάζουν τα πράγματα που συμβαίνουν και οι καθηγητέ θα πρέπει να του βοηθήσουν να καταλάβουν πώ μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα που του ενδιαφέρουν, πώ μπορούν να εμπλακούν ενεργά στην πολιτική. Με αυτή την κατανόηση θα έρθει και η διάθεση να ασχοληθούν με τα ευρωπαϊκά πράγματα και να πάνε να ψηφίσουν και στις ε, ευρωεκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι πολύ περίπλοκη ιστορία και εγώ όταν γεννήθηκε δεν ήμουν εκεί για την... και δεν ισχυρίζομαι την καταλαβαίνω πλήρω. Πώ θα υποστηρίξει κάτι που δεν καταλαβαίνει. Αν δεν ξέρει πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί όπω όπω ε, και θα προσπαθούμε όπως όπως να κρατήσουμε ζωντανή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ε, δημιουργήθηκε πριν από 60 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει φυγόκεντρες τάσεις και μέσω αυτής της εκπαίδευσης της αγωγής του πολίτη θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να την καταλάβουν πάλι. Ποιος ξεκινάει? Ο Τζόρτζ. Δεν θα και τόσο Κουλ, ε, στην απαντηθώ στην ε, Κιβοβό, είμαι μεγαλύτερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι αρκετά ηλικιωμένο στην πραγματικότητα. Οπότε έχω διαφορετική οπτική. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι είμαι υπέρ του να υπάρχει ανατροφοδότηση από οποιαδήποτε ηλικία. Φυσικά είναι, έχουν πάντα καινοτόμε ιδέε, όμω το κέντρο βαρύτητα είναι σε αυτού που είναι πάνω από 60. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και με τη βιοτεχνολογία. Θα μπορούν να ζουν άνθρωποι μέχρι τα 130 τους χρόνια. Άνθρωποι που τώρα είναι στην ηλικία σου. Όταν θα φτάσει στα 50-60 θα το καταλάβεις. Θα καταλάβεις όλο αυτό που λέω. Έκανες λόγο για ποικιλομορφία και η ποικιλομορφία στην ηλικία, στα ηλικιακά γκρου πρέπει να είναι και αυτό είναι ένα κομμάτι από αυτό που προτείνεις. Υπάρχουν ε, κοινωνιολογικές μελέτες που λένε ότι η ποικιλομορφία μειώνει την εμπιστοσύνη. Περιμένω μια ισχυρή αντίδραση από εσένα σε αυτό. Μερσέντες, Ρίτσαρντ, θα θέλετε να πάρετε το λόγο. Η Mercedes. Mm, molto, mm, molto brevemente. Πολύ σύντομα. Για την ανάγκη να γίνει μια πολύ πιο σοβαρή προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο αγωγής του πολίτη. Όλοι συμφωνούμε. Και πολύ περισσότερο το Κοινοβούλιο, το οποίο κατ' επανάληψη έχει πιέσει να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση μίλησε για προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα αγωγής του πολίτη. Συμφωνώ ότι είναι δύσκολο να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε ένα θεσμικό όργανο αν δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Άμα δεν, κα... δεν καταλαβαίνεις καν τα προβλήματα τότε. Άκουσα να, σας, να σταθώ και σε κάτι που είπατε προηγουμένως. Ότι πρέπει να γίνει πολλή προσπάθεια για τη, βελτια... για τη βελτίωση της online ε, διαβούλευσης. Που είναι ο κανόνας, αλλά που αφορά μόνο τα νομοθετικά κείμενα. Δεν θα αφορά τις πολιτικές, τις ε, αρχές, τις δράσεις και επομένως είναι κάτι το ψυχρό και δεν μπορεί ο απλός πολίτης, νέος ή λιγότερο νέος, να ενδιαφερθεί για ένα θέμα που στην πραγματικότητα είναι ιστορία, κλασική ιστορία των λόμπι. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις Επί ποιων θεμάτων μπορούμε να οργανώσουμε αυτές τις διαβουλεύσεις online, ούτω ώστε να καταστήσουμε πιο ενδιαφέρουσα την ανταλλαγή απόψεων. Πρέπει να δούμε κάποια μεγάλα θέματα που συνδέονται με τις πολιτικές, πριν από τα νομοθετικά κείμενα, τα οποία ενδεχομένω πρέπει να τροποποιήσουμε. Επ' αυτού έχετε να κάνετε κάποια πρόταση. Richard. Well, to liven things up, may I disagree with Θα διαφωνήσω με τον Τζόρτζ για την νεολαία. Δεν είμαι βέβαια στην ηλικία σου ακόμα. Πολλέ πολλές φορές ε, είναι παραπροχωμένη η απόψη μας. Είναι καλό να έχουμε μια φρέσκια ματιά στα πράγματα χωρίς προκαταλήψεις. Επίσης έχουμε εμπειρίες ε, και ξέρουμε πώς να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί, πώς να κινηθούμε οι νέοι. Πολλές φορές δεν έχουν αυτή τη γνώση και γι' αυτό χρειαζόμαστε μηχανισμούς να τους δώσουμε την ευκαιρία να εκφραστούν. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με τα πάντα, ε, με όλα όσα ακούμε. Είπατε κάτι ότι είναι τελετουργικές οι διαδικασίες. Πιστεύω ότι εφόσον είστε εσείς από την Μεγάλη Βρετανία να πείτε ότι εμείς ε, είμαστε πιστεύετε τελετουργικά, δείτε λιγάκι πώς είναι το Αγγλικό Κοινοβούλιο, εκεί και αν δεν υπάρχουν ε, τελετουργίες, εμείς είμαστε πιο πρακτικοί και εστιάζουμε στο διάλογο και στα αποτελέσματα. Αλλά το, να τα ακούω αυτό από εσάς μου φαίνεται περίεργο. Από την άλλη όμως ε, με προβληματίζετε και σκέφτομαι ότι θα πρέπει να το δούμε το θέμα. Θέλω και εγώ να μιλήσω. Είχαμε 3,5 αντιδράσεις από τους ευρωβουλευτές. Συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι συμμετοχική η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους περιλαμβάνει όλους. Όταν μιλάμε όμως για ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ε, ε, μιλάμε για τα δικαιώματα των πολιτών, όμως δεν μιλάμε για τις υποχρεώσεις τους. Και ειδικά μετά το δημοψήφισμα, ποια είναι η ευθύνη των πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης. Και τώρα λόγω σε εσά και πάλι, Ποιο θα μιλήσει πρώτος, ο Λεωνί. Ε, δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό που είπα για το τελετουργικό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα πρωτόκολλα και μη αναγκαίε δομέ. Πρέπει να δούμε τα πρακτικά θέματα, όπω είπατε και εσείς. Με απογοητεύει αυτό που άκουσα για την εμπιστοσύνη και για την ποικιλομορφία, πιστεύω ότι η ποικιλομορφία βοηθάει πάρα πολύ στο να ακουστούν οι απόψει των ατόμων στην κοινωνία και αυτό ε, είναι, αυτή η ουσία του ευρωπαϊκού κινήματο. Έχω αίσθηση προ αυτό που είπατε λοιπόν. Το να δίνουμε βήμα στου νέου ε, και παρέχοντα του πληροφορίε με πιο εύκολη ορολογία βοηθάει αυτό όμως που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι να ε, μπλέξουμε ενεργά τους νέους στη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω προτάσεις για συγκεκριμένα ονόματα, για κάποια θέματα, για το ονομάστε θέματα συγκεκριμένα σε πολλά πράγματα σπουδών, σχολείων πρέπει να εντάξουμε τέτοια θέματα γιατί ποτέ δεν μιλάμε ουσιαστικά για την ε, συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθε. Πολλοί δάσκαλοι φοβούνται να μας δείξουν τη δικιά τους πολιτική τοποθέτηση κάτι που δεν επιτρέπεται και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για βέλτιστες πρακτικές ώστε οι δάσκαλοι να μπορούν να βελτιώσουν την συμμετοχή και να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να α, συμμετέχουν και όσον αφορά τις ευθύνες που αναφέρεται. Άμα δείξουμε στα παιδιά πώς θα μπορούν να είναι ενεργοί πολιτικά, θα ε, μπορούν ε, στη συνέχεια, γιατί το βλέπω και με τον ε, εαυτό μου και με τους φίλους μας, ότι όταν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα και συμμετέχουμε, τότε είμαστε και έτοιμοι να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο που είναι η συμμετοχή της νεολαίας στην πολιτική ζωή. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα για όλους μας, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι ε, ακούμε πολύ συχνά ότι οι ναι, νέοι δεν χρειάζονται την πολιτική στήριξη γιατί η τεχνολογία είναι αρκετή για αυτούς. Θα ήθελα να ενημερώσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους που ήρθαν τώρα ότι θα πρέπει να απαντήσουμε μέσα σε ένα λεπτό. Αν θέλει να πάρει το λόγο, λοιπόν, να σας το δηλώσει. Ο Νίκολας, ο λόγος σε σένα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας προτείνω να αρχίσουμε να ψηφίσουμε νωρίτερα, στο 16, σε όλες τις εκλογές, για να, να βελτιώσουμε τη συμμετοχή στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε. Αυτή η ιδέα κυκλοφορεί εδώ και καιρό, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οι νέοι το θέλουν αυτό έντονα. Γι' αυτό το προτείνουμε όσο πιο συχνά γίνεται. Εγώ είμαι Αυστριακός όπου πριν από λίγα χρόνια κατεβάσαμε το όριο ηλικία. Και από πείρα σας λέω ότι πραγματικά βοηθάει τους νέους να κινητοποιηθούν πολιτικά. Αν κοιτάξετε τις φιγμομετρήσει, συχνά οι νέοι πιστεύουν περισσότερο στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που αισθάνονται τμήμα αυτής της ε, διαδικασία. Και όμως στην πραγματικότητα οι γνώμε του, ε, επειδή δεν έχουν πολιτική επιρροή, σπάνια ακούγονται το, να τους δώσουμε το πιο βασικό εργαλείο δημοκρατικής εμπλοκής στο δικαίωμα ψήφου είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά, ίσως πιο φιλικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση α, εκλογικά αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη σε αυτό για τον Brexit. Εάν μειώσουμε το όριο ηλικία στα 16, θα μάθουν οι νέοι να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία πολύ νωρίτερα και θα υποφεληθεί η δημοκρατική διαδικασία. Εάν ε, συμμετέχουν με περισσότερα ποσοστά, με μεγαλύτερα ποσοστά οι ευρωπαϊκοί οι νέοι στις ε, πολιτικές διαδικασίες, θα έχουμε πιο βιώσιμες πολιτικές, ε, θα προάγουμε θέματα που είναι πολύ πιο σημαντικά για τους νέους, για τα προβλήματα που αφορούν και απασχολούν τους νέους ε, και θα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις εκλογές. Φυσικά αυτό θα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και καλό θα ήταν να συνδυαστεί με αυτή την προσπάθεια ε, δραστηριοποίησης των πολιτών ε, μέσω της αγωγής του πολίτη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η η υποεκπροσώπηση των νέων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμποδίζει τη δημοκρατία μας. Η ιδέα μου είναι όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη να δεσμευτούν πολιτικά, ούτω ώστε να έχουν ποσοστώσει για του νέου σε όλε τι εκλογέ, από τι τοπικέ μέχρι τι ευρωπαϊκέ. Και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από τις ευρωεκλογέ του 19. Σ ε, κοιτάξτε, σε όλες τις εκλογές χρησιμοποιούνται ποσοστώσεις για τις γυναίκες. Αυτό είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις ε, για την εκπροσώπηση των γυναικών. Θα πρέπει τον ίδιο μηχανισμό ε, να εφαρμόσουμε τόσο ώστε να αυξήσουμε τον αριθμό των νέων πολιτικών. Ε, Ακούστηκε αυτή η ιδέα και υπάρχει ευρεία, ευρεία υποστήριξη αυτής της ιδέας. Όλα, αν δεσμευτούν όλα τα πολιτικά κόμματα για τέτοιες ποσοστώσεις, ε, θα θεωρούμαστε ότι έχουμε ίδια δικαιώματα, είμαστε εξίσου πολίτες και θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία. Και θα σταματήσει ε, η παραποίηση της εικόνας των νέων. Θα ε, δραστηριοποιηθούν περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Εάν είσαστε σοβαροί, μπορείτε να πάτε και παραπέρα από τις ποσοστώσεις. Ο Ρίμπαν Μαρί, ε, Γάλλος καθηγητής, είπε ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπο, υπερεκπροσωπούνται οι ηλικιωμένοι άσπροι άντρες. Θα πρέπει δηλαδή να σταματήσουν να υπερεκπροσωπούνται αυτή, αυτή η ηλικιακή κατηγορία για να στρεβλώνουν ας πούμε την κουλτούρα της πολιτικής. Θα πρέπει να αξιοποιείται η συμμετοχή των νέων. Είναι ε, εργαλείο και είναι και προϋπόθεση για μια πραγματική δημοκρατία. George, θες πάλι να πεις κάτι το προκλητικό και εγώ είμαι έτοιμη, λέει Σέι. Κοιτάξτε, εγώ θα συνεχίσω να σας απαντάω. Ε, το κάνω με ευγένεια, ας πούμε, και σεβασμό. Ξέρω ότι τα βρετανικά ήθη έχουν αλλάξει. Καταρχάς, για την ψήφο για τους νέους. Ε, αυτό που είπε ο αυστριακός εκπρόσωπος, ο κ. Σέρλιγκερ. Α, κοιτάξτε τα στοιχεία. Πολύ προσεκτικά. Υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση, όχι μόνο των νέων, αλλά ενός σημαντικού τμήματος των νέων, 25 με 30% είναι μια τάση, ας πούμε, ε, αντίδρασης κατά του κατεστημένου. Και μιλάμε ε, για μια υποστήριξη από μέρους τους των ακροαριστερών ή ακροδεξιών κομμάτων που δεν είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επομένως, προσοχή ε, για το τι εύχεστε, έτσι. Τώρα, για τις ποσοστώσεις για τους νέους, γιατί όχι. Αλλά γιατί να ξεκινήσουμε με τους νέους, γιατί τότε να μην σκεφτούμε δεκάδες άλλες ομάδες. Ας πούμε οι ανάπηροι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί όχι. Επίση, οι αριστερόχειρε. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με ποσοστό για αριστερόχειρε, Φερρυπίν. Uh, uh, <laughs> uh, εμείς στηρίζουμε την ψήφο στα 16, εμείς από τους εργατικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μακάρι να ήταν να ίσχυε αυτό στο δημοψήφισμα, γιατί θα είχε γύρει αλλού η πλάστικα. Τώρα για τις ποσοστώσεις και την ιδέα αυτή. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε γι' αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Διότι την αρμοδιότητα την έχει η εθνική νομοθετική πρωτοβουλία. Ο σωστό τρόπος να το επιτύχουμε αυτό είναι εσείς να ασκήσετε πίεση στα ε, κόμματά σας και στην ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Η προσέγγιση σας όμως είναι η σωστή. Last MEP. Η κυρία Σπινέλη παρακαλώ. Είναι η τελευταία που θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Μα, ε, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένη στη συνάντηση αυτή. Αλλά δεν συμφωνώ με αυτά που είπε και ο κ. Σέπφλιν για την κομβική σημασία και τον κομβικό ρόλο που παίζουν οι ηλικιωμένοι πάνω από 60 δηλαδή. Και το λέω εγώ που είμαι και μεγαλύτερη, πιο ηλικιωμένη από εσά. Γιατί η Ευρώπη που οικοδομούμε, ναι, ναι, νομίζω ότι είμαι πιο μεγάλη από εσά. Ναι, γιατί η Ευρώπη που χτίζουμε, αυτοί που θα τη ζήσουν το πετσί τους κυρίους, δεν θα είναι κυρίως οι νέοι και πολύ περισσότερο, για πολύ περισσότερο χρόνο, αλλά και οι επόμενες γενιές. Αυτοί θα είναι οι μελλοντικοί κυβερνήτες, οι μελλοντικοί ηγέτες. Είμαι πολύ θερμός υπέρμαχος του να μειωθεί το όριο ηλικίας για τις, τη συμμετοχή εκλογές. Επίσης, αυτή την επιτροπή έχουμε συζητήσει μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για την ηλεκτρονική δημοκρατία. Ο εισηγητής είναι παρόν. Είναι ο συνάδελφος που κάθεται μπροστά μου. Και απευθύνεται κυρίως στους μελλοντικούς ηγέτες. Ένα άλλο βασικό εργαλείο είναι αυτή η πρωτοβουλία για τους πολίτες. Επ' αυτού, ο κ. Σέφλιν πρότεινε και μια θαυμάσια μεταρρύθμιση, την οποία δεν δέχτηκε ακόμα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα εργαλείο, ένα ακόμα εργαλείο, από το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε και το οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε. Ο Νικόλαος ένα λεπτό και η ΣΕΙ επίσης. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Σέπλιν και στα λεγόμενά του. Να συμφωνήσω ότι οι νέοι ριζοσπαστικοποιούνται κάπως. Όμως, δύο είναι οι δρόμοι μας. Δύο τρόπους έχουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αυτό που προτείνετε εσείς είναι να συνεχίσουμε να εγκαταλείπουμε τους νέους. Είναι αυτός ο ένας δρόμος. Αν δεν τους αφήνουμε να, ψηφίζουμε, να ψηφίζουν γιατί είναι εξαιρετικά ριζοσπαστικοί στη στάση τους, ουσιαστικά συνεχίζουμε να τους εγκαταλείπουμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Ο άλλος δρόμος είναι να τους εμπλέξουμε στη διαδικασία να τους κάνουμε να συμμετάσχουν στην διαδικασία. Θα πρέπει για να απορριζοσπαστικοποιηθούν να τους δώσουμε το δικαίωμα να αποτελέσουν μέρος της πολιτικής διαδικασίας. Και πολύ συχνά τα πολύ ριζοσπαστικά κόμματα είναι αυτά τα οποία ε, ε, αφού γράζονται καλύτερα τους νέους δυστυχώς. Θα πρέπει και τα κόμματα του μεσαίου χώρου να δώσουν περισσότερη σημασία ε, στα ζητήματα των νέων. Μπορώ να απαντήσω εν συντομία, λέει ο κύριος Βουλευτής. Είμαι απολύτως υπέρ του ορίου ηλικία στα 16. Όμως, στα 16 απλά σε δύο χρόνια νωρίτερα, εάν έχεις το δικαίωμα να ψηφίσεις. Πολλές και διαφορετικές απόψεις θα ακούσουμε, λέει η Πρόεδρος, εάν ρωτήσουμε τον, το καθένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεχωριστά. Εισέγει. Κύριε Σαπλίν, καταρχά να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, Σα σας σέβομαι και σας τιμώ. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι ποσοστό αυτές είναι ίδιε με αυτέ που αναφέρετε. Για παράδειγμα, ε, αυτό το οποίο λειτουργεί πολύ καλά σε σχέση με τους Ινδούς, για παράδειγμα, είναι ότι κοιτάζουμε σε κάθε συμβούλιο να έχουμε και έναν εκπρόσωπο της, αυτής της κοινότητας ή της εκάστοτε κοινότητας και νομίζω ότι αυτά λειτουργούν όλα πολύ καλά. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε όσο να τον καλύτερη αντιπροσώπευση της κοινωνίας. Κύριε Κόρμπετ, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ελπίζω να υπάρξει πολιτική δέσμευση, υπόσχεση για να έχουμε περισσότερους νέους πολιτικούς, περισσότερους νέους βουλευτές και εδώ και στο, σε εθνικό επίπεδο. Και συμφωνώ απολύτως. Το Βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστημα είναι απολύτω τελετουργικό στι εναρκτήριε ομιλίε, δίνει υπερβολικά μεγάλη σημασία στο πρωτόκολλο. Αν ρωτήσετε τους νέους, θα δείτε ότι τους συνεπέρνουν τα μεγάλα ζητήματα. Όμως στη διαδικασία δεν βρίσκουν τίποτα στο οποίο να μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους λόγω ακριβώς ε, του, αυτής της πολύ τυπικής, υπερβολικά τύπολατρικής διαδικασίας. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα δούμε κατά πόσο τα μηνύματα θα παραμείνουν ίδια από τη νέα γενιά. Ξέρετε, αποκομίζω την αίσθηση ότι συχνά δεν συνειδητοποιούμε αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα στις μελέτες. Ότι δηλαδή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αλλά και αλλού, την πρώτη φορά που ψηφίζει ένας νέος, συνήθως ψηφίζει ένα πολύ ακραίο κόμμα. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε, πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα, πρέπει να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα και αυτού του φαινομένου αλλά και του, του, πώς ψήφισε ο κόσμος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε ε, σε διαφορετικά κράτη-μέλη το ότι οι νέοι μοιράζονται περισσότερα κοινά με νέους από άλλα κρατημέλη. Δηλαδή, ανεξαρτήτως χώρας, η ομάδα αυτή παρουσιάζει πολύ κοινά χαρακτηριστικά και πολύ κοινέ ανάγκες και οφείλουμε πραγματικά να το λάβουμε αυτό υπόψη. Εδώ ολοκληρώνεται αυτή η ακρόαση. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Ε, για το ότι ήρθατε εδώ, για το ότι ακούσατε, για το ότι μιλήσατε. Κάποιες απόψεις δεν ακούστηκαν, κάποιες άλλες μπορέσαμε να τις ακούσουμε και ελπίζουμε να έχουμε και τους επόμενους αυτούς που θα πάρουν τη σκητάλη από εσάς του χρόνου στην αντίστοιχη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Εποθέσεων. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σε δύο λεπτά ε, συνεχίζεται η συνεδρίαση. Thank you very much. Thank you,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 Να συνεχίσουμε την ε, συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι. So we are now moving to point... Προχωράμε στο σημείο 8, στην μερίσια διάταξη. Ο Γκίφερ Χόφστατ που είναι μαζί μας σήμερα και θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για νέα τροπολογίες στην έκθεσή σας. Δεν πιστεύω να συζητήσετε την καθεμία μεμονωμένα, ωστόσο Έχεις όλο τον χρόνο στη διάθεσή σου και χωρίς να καθυστερούμε ας ξεκινήσουμε με τον Γκί ως εισηγητή. Θα είμαι πολύ σύντομος. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε όλες τις τροπολογίες. Θα παρουσιάσω κάποιες ε, συμβαστικές προτάσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις σε αυτές τις τροπολογίες. Ε, προετοιμάζω και εγώ με τους ε, δικούς μου ανθρώπους ένα, ε, ένα αριθμό συμβαστικών προτάσεων και η πρόθεσή μου είναι την επόμενη εβδομάδα να έχω μια συνεδρίαση με τους ε, σκιώδες από τις ε, ομάδες για να δούμε αυτές τις συμβαστικές ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματα που έχουν προκύψει. Η πρόθεσή μου είναι την επόμενη εβδομάδα να έχω συνεδρίαση με όλους τους ε, σκιώδες συγκητές από όλες τις ομάδες της ΑΦΚΟ με βάση αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Ένα στοιχείο που θέλω να, στο οποίο θέλω να εστιάσω και θα προσπαθήσω να το πλήσουμε με μία νέα πρόταση για αυτό το άρθρο. Είναι το άρθρο 10 της πρότασης και που αφορά την, το στάτους σύνδεσης. Είχα την αντίθεση πολλών συναδέλφων που θεωρούν ότι η πρόθεση είναι να διαχωρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύο τύπους κρατών μελών. Πλήρη μέλη και συνδεδεμένα μέλη. Δεν αφορά αυτό, όχι σε καμιά περίπτωση. Η ιδέα είναι δεν αφορά τα τρέχοντα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε τα μελλοντικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά τις χώρες που δεν θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που δεν επιτρέπεται ενδεχομένω. θα πρέπει να το αναλογιστούμε αυτό το θέμα, γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα, ήδη σήμερα, και θα είναι και πιο προφανές μετά τις ε, επιτυχημένες διαπραγματεύσεις για το Brexit, για κάθε χώρα ή κάθε κράτος θα έχουμε ένα διαφορετικό ε, μοντέλο Έχουμε την περίπτωση της Νορβηγίας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Έχουμε άλλη περίπτωση με την Ελβετία και άλλη περίπτωση, άλλο καθεστώ με την Νορβηγία. Είναι διαφορετικέ περιπτώσει, διαφορετικού είδου συμφωνίε. Και με την Τουρκία είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε τελωνιακή ένωση και με την Ουκρανία. Άλλου είδου ε, ε, συμφωνία. Συμφωνία σύνδεση με τον στόχο ε, περισσότερη περαιτέρω ενσωμάτωση. Ισλανδία, άλλη κατηγορία κι αυτή. Όπως και η Ισλανδία. Και πάει λέγοντας. Θεωρώ ότι έχουμε τουλάχιστον έλλειψης έννοιων. εντός της ενός, αλλά ακόμα την έλλειψη εκτός. Έχουμε ένα μπάλωμα ουσιαστικά, ένα... μια σειραφή. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το άρθρο 10, προτείνω αντί να έχουμε 6, 7, 8, 9 διαφορετικούς τύπους συμφωνιών, εταιρικών σχέσεων, θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε, με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επανέλθουμε ε, στην ιδέα των ιδρυτικών πατέρων, μια ιδέα του 53, ότι Έχουμε τα μέλη και μετά οι υπόλοιποι περιλαμβάνονται σε εταιρικέ σχέσεις. Και αυτές οι εταιρικέ σχέσεις πρέπει να ε, περιλαμβάνουν και μια σειρά όρων. Να εφαρμόζεται το κράτος δικαίου, παραδείγματος χάρη και η εξή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η γενική ιδέα. Ήθελα να το αναφέρω γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποια, κάποιοι βουλευτές από χώρες που θεωρούν ότι αυτό το στάτους σύνδεσης είναι ένας τρόπος για να απομακρύνουμε κάποια μέλη. Ενώ είναι το αντίθετο ακριβώς. Όπω είπα και πριν, θα προτείνω μια, μια καινούργια διατύπωση στου σχεδόν συγκητέ την άλλη εβδομάδα για το άρθρο 10 και για άλλα άρθρα για να άρουμε αυτή την παρεξήγηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το κείμενο που έχουμε προτείνει. Okay. Thank Ευχαριστώ, Παύλο Ράντζο, για το EPP, για το ΕΛΚ. Καταρχάς ήθελα να πω ότι ότι έχουμε ένα περίπλοκο σύνολο τροπολογιών και πολύπλοκες είναι επίσης και οι συμβαστικές προτάσεις που θα πρέπει να τις προσέξουμε πολύ. Θεωρώ ότι είναι πρόωρο, πρόημο το στάδιο για να έχουμε μια πολύ σταθερή και πάγια άποψη για το τελικό ε, μας έργο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να τονίσω δύο κέρια ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι κατά κάποιο τρόπο οι τροπολογίες περιλαμβάνουν ε, μια πολύ έγκυρη ανησυχία γιατί όταν μιλάμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας υπόψη την ανάγκη μεταρρύθμισης, μετατροπής της συνθήκης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολύ συγκεκριμένες λύσεις, αλλά ακόμα περισσότερο να δούμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θέλουμε να γίνουν οι μετατροπές και να εντοπίσουμε τον ενδειγμένο δρόμο για τη λύση, αλλά όχι μια συγκεκριμένη λύση. Δεν σχεδιάζουμε λοιπόν μια νέα συνθήκη σε αυτή την έκθεση, αλλά εντοπίζουμε ποιοι είναι οι τομεί και ποια είναι η κατεύθυνση σε κάθε τομέα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε ευρεία ομοφωνία. Αν όμως μπούμε σε λεπτομέρειες και επειδή ο καθένας μας δεν έχει μόνο όνειρα για την Ευρώπη αλλά και συγκεκριμένα συγκεκριμένε ιδέε, θα μπορούσαμε να περάσουμε στη συνέχεια στι λεπτομέρειε. Αυτό θα βοηθούσε και τον εισηγητή και τους σκιώδει εισηγητή να πετύχουν ε, μια ε, λογική συμβαστική πρόταση. Μια δεύτερη παρατήρηση σχετικά με αυτό που έθιξε ο Γκί για το στάτους σύνδεσης, καθεστώς σύνδεσης. Είμαι πολύ ανοιχτόμυαλος και πρόθυμος ακόμα να αλλάξω και την άποψή μου. Γιατί θα πρέπει φυσικά να διαβουλευθώ και με το ΕΛΚ, να μάθω ποιες είναι οι απόψεις εκεί. γιατί υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι από τη μία καταλαβαίνω την έννοια του καθεστώτου σύνδεσης, κατάλαβα από την αρχή ποια ήταν η πρόθεσή σας για αυτούς που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως από την άλλη δεν βλέπω πώς θα λειτουργήσει αυτό το καθεστώ σύνδεσης. Γιατί έχουμε την Τουρκία, έχουμε και την Νορβηγία. Και επομένω, αν κάνουμε λόγο για κράτη που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως θα πρέπει να έχουμε ευελιξία για να δούμε διαφορετικούς, ε, διαφορετικές συνθήκες και τα διαφορετικά την κάθε περίπτωση μονομένα του κάθε κράτους. Φυσικά θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια, όπως το κράτος δικαίου, την, ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως προς αυτά συμφωνώ όσον αφορά στο θεσμικό σχεδιασμό του κράτους που θα είναι σε καθεστώς σύνδεσης, το να είναι μονάχα ένα το καθεστώς σύνδεσης, που θα ισχύει για όλα τα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ ότι αυτό δεν ε, είναι λογικό. γιατί άλλη σχέση θα έχουμε με την Ορβηγία, με, την, ε, με το Ρωμανό Βασίλειο, με την ε, Ελβετία ε, και άλλοι με την Τουρκία, με την Ουκρανία κτλ. Αλλά δεν θέλω ότι υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Μια δεύτερη παρατήρηση γιατί ότι πολλοί έχουν μπερδέψει δύο πράγματα. Το τι θα κάνουμε με τα κράτη που είναι ήδη εντό τη Ένωσης, γιατί μία από τι ε, ανησυχιε που θίγεται στο πρώτο σχέδιο είναι ότι ε, έχουμε μία πολύ ασύμετρη Ένωση, γιατί κάθε κράτο έχει άλλου είδου ε, συμμετοχή, άλλο πράγμα είναι η Δανία, άλλο η Ιρλανδία κτλ. Κάθε κράτος μέλος έχει άλλου είδους σχέση και βαθμό συμμετοχής. Προσπαθώ να υπερασπιστώ και την δικιά μου άποψη, αλλά να δω τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνω μια ιδεοθύελα ότι αν έχουμε δύο είδη σύνδεσης, δύο είδη, δύο καταθεστώτα ε, συμμετοχής, αυτά που συμμετέχουν στη ζώνη Σέγγεν, στην Ευρωζώνη κτλ. και τα άλλα κράτη που θέλει στην νέα αγορά κτλ. κτλ. Ίσως θα μπορούσαμε έτσι να τα κατηγοριοποιήσουμε, ίσως θα μπορούσε αυτή να είναι μια ενδεδειγμένη λύση. Αλλά βλέπω σε πολλές τροπολογίες μια διαφορετική αντίληψη ότι πρέπει να έχουμε ένα καθεστώς και να ζούμε με αυτή την ε, ποικιλομορφία, να ανεχτούμε αυτή την ποικιλομορφία, γιατί έχουμε 19 κράτη στην Ευρωζώνη και τα υπόλοιπα έχουν δεσμευτεί ότι θα εισέλθουν επίσης. Επίσης το ίδιο και με την ε, ζώνη Σέγγεν. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη φτάνουν σε έναν τελικό βαθμό ενσωμάτωσης, άρα θα πρέπει να σκεφτούμε ε, και να προτείνουμε αυτό, αυτή την πρόταση για συμμετοχή με δύο διαφορετικά καθεστώτα. Θεωρώ ότι λοιπόν αυτό δημιουργεί έναν ε, διχασμό όχι ως προς την ιδεολογική προσέγγιση, αλλά βλέπουμε ότι οι βουλευτές από το ίδιο κόμμα και από την ίδια χώρα έχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτή είναι η εμπειρία μου από τις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να οριμάσει λίγο η σκέψη το καλύτερο θα ήταν να εστιάσουμε στην δεύτερη τάση, να επιτρέψουμε δηλαδή κάποιο είδος ασύμμετρης ε, γεωμετρίας όπου θα έχουμε ε, ειδικές συνθήκες για κάποια κράτη-μέλη. Αυτή βλέπω την τάση που προτείνεται στις τροπολογίες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτή τη συζήτηση πρέπει να την έχουμε με τους σκιώδεις συζητητές, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αντίκτυπος που θα έχουν στον σχεδιασμό των συμβαστικών προτάσεων, στην οικονομική διακυβέρνηση επίσης, στην αμυντική ένωση θέματα μετανάστευσης κτλ. Αυτή είναι λοιπόν η άποψή μου. Πρέπει να κάτσουμε όμως γύρω από ένα τραπέζι και να ε, συζητήσουμε, να παρουσιάσουμε τις ιδέες μας και να παρουσιάσουμε στη συνέχεια εδώ στην Επιτροπή μια πιο πάγια άποψη. Γιατί χρειάζεται ακόμα να το σκεφτούμε το θέμα. Ευχαριστώ, Πασκάλ.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 de cette question institutionnelle les questions plus de gestion. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir donné la parole maintenant. Yeah, for large we support the Verhofstadt draft report. I think it is really forward-looking. It is inspiring, giving ideas how we could have more unity instead of more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 Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ισορροπία στην εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης στα θεσμικά όργανα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και τούμπαλιν. Να επαναλάβω αυτό που είπα πριν από λίγες εβδομάδες. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Φερχόφσταντ επικεντρώνονται στην εμπιστοσύνη προ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Από την άλλη πρέπει να καταπολεμήσουμε την κρίση και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα, αμοιβαίο, ή μάλλον ένα σύστημα αμοιβαία εμπιστοσύνη που σέβεται την ποικιλομορφία. Έχω τελείως διαφορετική ιδέα και ιδεολογία και προσέγγιση και ίσω και διαφορετικού στόχου. Δεν θα ξεκινούσα από μια επίσημη αλλαγή των συνθήκων θα ξεκινούσα από τη διοργάνωση μιας πανευρωπαϊκής συζήτησης για αυτό το θέμα. E, Χωρίς ε, τελεολογικό σκοπό στη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Ροζιέ από το ΕΛΚ που ζήτησε σύνεση. Είναι μια πολύ λεπτομερής έκθεση αυτή. Έχει πολύ συγκεκριμένες συστάσεις μείωση της εξουσίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, να σταματήσει να έχει εξουσία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Φερρυπίν. Όλες αυτές οι αποφάσεις μπορεί να γίνουν, αλλά στο τέλος της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων και όχι εξ Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίσει να εργάζεται επί αλλαγών στις συνθήκες, τότε θα πρέπει να καλέσει τον κόσμο να συμμετάσχει, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικό και ισορροπημένο στην προσέγγιση του. Δεν θα πρέπει να είναι μονόπαντο. Και θέλω λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, να συνταχθώ με τον κύριο Χωζέ που ζήτησε προσοχή και επίσης και μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία ε, αλλαγής ε, των συνθήκων. Η κυρία Μπάρμπαρα Σπινέλη είναι η επόμενη μιλήτρια. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσής του και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τους συμβασμούς. Να πω από την αρχή ότι υπάρχουν κάποια τμήματα που μου αρέσουν για την εσωτερική ασφάλεια, η οποία δεν θα πρέπει να γίνει πρόσχημα για να αποφύγουμε πιο θαραλέες πολιτικές ε, ασύλου και ένταξης, για να περάσει η εξωτερική πολιτική στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στην κοινωτική μέθοδο που θα πρέπει να πριτανεύει έναντι της ε, διακυβερνητικής μεθόδου, επίσης συγκεκριμένα δικαιώματα στο Ευρωκοινοβούλιο, ξεκινώντας από το δικαίωμα προ νομοθετικής πρωτοβουλίας και το δικαίωμα έρευνας, σύστασης ερευνητικής επιτροπής. Συμφωνώ και με αυτό που είπατε για την ΕΚΤ που να είναι ο δανειστής ίστατη της καταφυγής, όπως είπα και σε προηγούμενε συνεδριάσεις, έχω μια σειρά από αμφιβολίε που τις εκφράζω μέσω τροπολογιών. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω μερικές, ε, αλλά με συνοπτικό τρόπο. Καταρχάς, έχω επιφυλάξεις αρκετά έντονες για το προήμιο για την αιτιολογική σκέψη, δηλαδή που δικαιολογούν και διάφορα ε, κατοπινά σημεία του ψηφίσματος. Αυτό που μου λείπει πάρα πολύ είναι μια κριτική και αυτοκριτική ανάλυση για την κρίση που μας δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατά τη γνώμη μου έφτασε στο πικ κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για την Ελλάδα και οδήγησε μοιραία στο Brexit. Νομίζω ότι αυτά τα δύο γεγονότα Τη Ελλάδα και τη Βρετανία που να συνδεθούν. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο όχι μόνο γιατί τα θεσμικά όργανα λειτουργούν άσχημα, δεν συντονίζονται καλά κτλ. ή δεν είναι αρκετά ομοσπονδιακά. Ο, η ομοσπονδιακότητα έχει νόημα αν υπάρχει μια αλληλέγγυα κοινότητα. Αν υιοθετούν πολιτικές που δεν διαιρούν τις κοινωνίες μας και δεν δημιουργούν όλο και περισσότερη αηδία προς την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ο φεντεραλισμός δεν είναι μια τεχνική και δεν αρκεί από μόνος του για να ξαναδώσει στους Ευρωπαίους πολίτες την εμπιστοσύνη που έχασαν και την αισιοτικά που ανήκουν. Ούτε με πείθει ανάλυση για την κρίση, η πολυκρίση όπως λέει η έκθεση του Φερχόφσταντ. Κατά την άποψή μου, η κρίση είναι της Ευρώπης δεν είναι κρίση που αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε, που δίνουμε απαντήσεις στην κρίση, αλλά δεν υπάρχει κρίση της μετανάστευσης, αλλά κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε μεταναστευτικές ροές και ροές προσφύγων, που αυτή τη στιγμή είναι το 0,2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Δεν υπάρχει μόνο κρίση χρέους, αλλά κρίση χωρών που επίσης επειδή είναι σε πλεόνασμα, σε πλεονασματική κατάσταση δεν επεκτείνουν την οικονομία τους. Όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργο Λάινεν, τα εθνικά κοινοβούλια συχνά δεν έχουν την εξουσία, τη δύναμη, τη δυνατότητα να παρακολουθούν πραγματικά αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις και να ελέγχουν αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις τους. Έχω την αίσθηση ότι η έκθεση δικαιολογεί πολιτικές οι οποίες δεν λειτουργούν καλά και που απέτυχαν ποικιλοτρόπως. Δεν αρκεί να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε έναν άνευ προηγουμένου σκεπτικισμό, μια επιστροφή του εθνικισμού, χωρίς να αναφέρουμε ποιες είναι οι λανθασμένες πολιτικές που προκάλεσαν και εξακολουθούν να προκαλούν εκτεταμένη δυσπιστία. Πάω τώρα στις ε, τροπολογίες επί του διατακτικού και αναφέρω μόνο τις πιο σημαντικές. Από το πρώτο άρθρο ζητάτε μία, ένα εξυγχρονισμό της διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν πάτε όμως στην ουσία της κρίσης, την ε, θεαματική έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, το ότι δεν υπάρχουν πια κάποια δικαιώματα, τα οποία αναφέρουν διάφορα άρθρα της συνθήκης, όπως το 2, 3, 6, 11 δεν υπάρχει μία ε, πολιτική στην Ευρώπη εξισορρόπηση των διαφορών ε, κέντρων εξουσίας. Άρθρο 13, όπου λέτε ότι δεν υπάρχει σύγκληση και ανταγωνιστικότητα και την καταγγέλλετε αυτή την έλλειψη. Αυτό που μου λείπει εδώ είναι να αναφέρετε τις κοινωνικές ανισότητες και να αναφέρετε την ε, αποδυνάμωση των πολιτών, που είναι η πραγματική λόγοι για αυτό το κύμα δυσπιστίας απέναντι στην Ευρώπη. Στο 14 Λέτε πολύ σωστά ότι ούτε το ε, Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ούτε η ρήτρα για το bailout έδωσαν τις ε, προβλεπόμενες λύσεις. Αλλά όμως δεν κάνετε τις κριτικές που ακούγονται τόσες πολλές από πολλούς πολίτες για τις συνταγές ε, λιτότητας, όχι μόνο από τους πολίτες, αλλά και από το δουνού του. Αν διάβασα σωστά την ε, έκθεση, μιλάτε για τις πολλές παραβιάσεις απέναντι στο σύμφωνο. Νομίζω ότι υπάρχει μία διαγνωστική καθυστέρηση σε σχέση με αυτό που λένε σε άλλους χώρους εδώ. Λυπάμαι επίσης που δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στην ε, πρόταση για ένα νέο ευρωπαϊκό deal, για ένα new deal. Ε, στο άρθρο 13 εγώ προτείνω κάτι, αλλά υπάρχουν πολλές ιδέες. Να ε, χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από νέους ίδιους πόρους που θα τροφοδοτούνται από ένα κοινό φόρο κληρονομιάς, ένα φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ένα φόρο επί των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Άλλη πρόταση είναι η Ένωση να προσυπογράψει την κοινωνική χάρτα και η συμπερίληψη των κριτηρίων της χάρτας στον ορισμό, στον, στις διάφορες οικονομικές πολιτικές. Σε ό,τι αφορά την έκθεση των πέντε προέδρων, ε, σημείο ή e, άρθρο 16, εσείς συμφωνείτε εν μέρη, εγώ, εγώ συμφωνώ ακόμα λιγότερο. Στην τροπολογία μου κάνω μία κριτική για την έκθεση και, από, και για τις λεγόμενες διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, που βασίζονται μόνο σε ανταγωνιστικότητα, που ως βασικό στόχο έχουν την αδιάρθρωση της αγοράς εργασίας και την εξίσωση προς τα κάτω των μισθών. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η συνταγή για να βγούμε από την κρίση και την ύφεση. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορώ να δεχτώ την πρόταση αυτή που σε άλλους καιρούς και με άλλες πολιτικές θα ήταν πολύ θετική να υπάρξει ένα κοινό Υπουργείο Οικονομίας ή Εξωτερικών με έναν Υπουργό Οικονομίας και ένα Υπουργό Εξωτερικών, γιατί υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβουμε τα λάθη του ευρώ. Δηλαδή, διάφορες ψευδεστήσεις ε, που θα μας δίνουν ε, την εντύπωση ότι αν φτάσουμε θεσμούς και θεσμικά όργανα, θα φτάσουμε ως εκθαύματος στην Πολιτική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μου πείτε ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός της ε, έκθεσης. Ούτε αυτός ε, της έκθεσης Μπροκ και Μπρέσο που μιλάτε για τις ε, συνταγματικές αναθεωρήσεις και όχι για τις πολιτικές ένωσης. Αλλά και στις δύο εκθέσεις συμφωνείτε με συγκεκριμένες πολιτικές. Και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο Πασκάλ Και αυτό εξηγεί το γιατί δεν μπορώ να συμφωνήσω με την έκθεση. Ότι εδώ δηλαδή μιλάμε μόνο, ότι πρέπει να μιλήσουμε σε αυτήν την έκθεση μόνο για θεσμικά θέματα, γιατί στην πραγματικότητα έμεσα γίνεται λόγος και για πολιτικά θέματα. Ευχαριστώ. Ε, ο Φάμπιο για το EDD η FDD, συγγνώμη, θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος. Θέλει να μιλήσει από το FDD. Το σκέφτηκα πολύ καιρό. Το θέμα με τις τροπολογίες στην πρόταση του κυρίου Φερχόφστατ. Όπως και με την πρόταση της κυρίας Μπρεσό και του κυρίου Μπρόκ. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι αδύνατο με την πρόταση του κύριου Φερχόφστατ. Δεν θα θέλει να ξοδέψει το χρόνο του σε τροπολογίε. έχουμε τόσο μεγάλε διαφορέ προ ε, την πρόταση αυτή που δεν μπορούν να συμβαστούν. Ε, ο κ. Φερχόφστατ ε, έχει τη δική του λογική. Θεωρώ ότι ε, θεωρεί ότι βρίσκεται, ένα ευρωπαϊκό, βρίσκεται μέσα στο ευρωπαϊκό τούνελ. Και το άρμα του είναι να μειώσει τη δύναμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όμως βρισκόμαστε στο πιλωτήριο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Υπάρχουν και εδώ πέρα μέσα στο Κοινοβούλιο πολλοί που είναι επικριτές του Ευρωπαϊκού Σχεδίου. Εδώ όλα φαίνονται απλά, αλλά αν δείτε απ' έξω τι συμβαίνει, έξω από το πιλωτήριο, τότε βλέπετε τα προβλήματα που υπάρχουν. Έχετε περιορισμένη όραση από το πιλωτήριο και όταν υπάρχουν προβλήματα αυτά οφείλονται στην αποτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με την ίδια λογικό είναι λογικό να ενισχύσουμε την περαιτέρω σωμάτωση, τη συνταγματική μεταρρύθμιση Και όλα αυτά δημιουργούν ε, στρεβλώσεις, όπως έχουμε δει στην Ευρωζώνη. Βλέπουμε ότι τρεις φορές την ημέρα παρακολουθούμε την ε, Ελλάδα, όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει μια νομισματική ένωση που δημιουργεί μια πολιτική σφαίρα που είναι αντιευρωπαϊκή. Και η λύση ποια είναι αντί να βρούμε έναν τρόπο να ε, έρθουμε πιο κοντά και να ενώσουμε τις ταυτότητές μας, είναι να πούμε ότι ε, έχουμε τις εθνικές ταυτότητες, ότι οπισθοδρομούμε η λογική δηλαδή ενός ηλικιωμένου ανθρώπου, ενός γέρου. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι διαφορετική η λύση. Ο 21ος αιώνας πρέπει να ε, μας δώσει την απάντηση σε αυτά τα θέματα περισσότερη ένωση, ευημερία, περισσότερη ασφάλεια, λιγότερη μετανάστευση. Δεν θα μπορέσει να τα παρέχει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα ο κύριος Τίμερμανς, που είναι τόσο ε, κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τόσο επικριτικός απέναντί της. Όταν ο ίδιος ο Τίμερμανς λέει ότι δεν είναι βέβαιο ότι όλα αυτά δεν θα οδηγήσουν στην καταστροφή και ότι είναι καιρός να πατήσουμε το φρένο. Και αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω και να πετύχω για την πρόταση της Μπρεσό και του Μπροκ, προτείνοντας τροπολογίες, ώστε να τους αποτρέψω από την πρόταση για αλλαγή της συνθήκης, μεταρρύθμιση. Η σταθερότητα μπορεί να μας παρέχει πολλά, όπως είπε και ο κύριος Τιμερμάνς, ε, στο ιστορικό σταυροδόμιο στο οποίο βρισκόμαστε, γιατί αν δεν ελέγξουμε την κατάσταση, τότε μπορούμε να τον χάσουμε πλήρως τον έλεγχο. Αν ακολουθήσουμε τη λογική του κυρίου Φερχόφστατ, θα αποσταθεροποιήσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μπορείτε να με κατηγορήσετε και να πείτε ότι ε, αυτό εξυπηρετεί δική μου λογική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, anybody, ε, we still have Max Anderson, please. Ο Max Anderson. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για το έργο του, προσπαθώντας να εξηγήσει με ακρίβεια αυτά που θέλει να πετύχει. Υπάρχουν κάποια σημεία που εκτιμώ ιδιαίτερα σε αυτή την πρόταση. Οι προτάσεις για να βρούμε λύσεις για κοινέ ευθύνε σε σχέση με τη μετανάστευση και για την επίλυση της κρίσης. Παράγραφη στο άρθρο 7. Αυτά είναι τα καλά στοιχεία της πρότασης. Όσον αφορά όμως την υπόλοιπη έκθεση, θεωρεί ότι παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Αν Αναρωτιέμαι, οι μελλοντικέ γενιές πολιτικών επιστημόνων θα... τι θα σκεφτούν για αυτή την έκθεση όταν θα την διαβάσουν στα βιβλία της ιστορίας θα μείνουν έκπληκτοι που τόσο σύντομα μετά από την απόφαση ένα από τα ιστορικά κρατημέλη να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μετά από αυτή την απόφαση, την ιστορική στιγμή ότι είναι τόσο συγκεντρωτική αυτή η πρόταση και τόσο φιλόδοξη και που προωθεί ένα πρόγραμμα, ένα project υπερκράτους θεωρώ ότι οι πολιτικοί επιστήμονες του μέλλοντος θα εκπλαγούν πραγματικά για αυτή την αντίδραση ενός μέρου της ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ότι είναι η πρόταση αυτού του σχεδίου. Αν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, τότε θα είναι κάτι πραγματικά επικίνδυνο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θύμα της συγκεντρωτικότητας δεν λειτουργεί η Ευρωζώνη, δεν είναι λειτουργική και δεν θα είναι λειτουργική για το προσεχές μέλλον. Το να προχωρήσουμε με περισσότερα, περισσότερα από τα ίδια μέτρα είναι πραγματικά επικίνδυνο. Περιορίστηκα σε 42 τροπολογίες, κάνοντας το διαχωρισμό ανάμεσα στην τοποθέτηση την κεντροαριστερή, την πραγματιστική τοποθέτηση της κεντροαριστεράς και την έκθεση του κ. Φερχόφστατ. Γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες και να μιλήσω για κάθε τροπολογία ξεχωριστά. Όμως θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι σαν να οδηγούμαστε στον γκρεμό. Αναμένω λοιπόν το διάλογο που θα έχουμε. Όμως θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα που είναι και το πιο σημαντικό. Η Σουηδία αποφάσισε ένα δημοψήφισμα ότι δεν θα γίνει μέρος της, μέρος δεν θα συμμετάσχει στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω με αυτή την ευκαιρία ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα ακολουθεί στο επερχόμενο μέλλον την ζώνη ήταν μια αποτυχία για τα κρατη και θα συνεχίσει να είναι αποτυχία για τα κρατημέλη μελη Είμαστε σε βαθιά ύφεση και φυσικά η Σουηδία δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτό και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σουηδίας και άλλες χώρες. Θα κρατηθούν μακριά από αυτό το ιδιαίτερα επικίνδυνο πείραμα. Έτσι θα έχουν τα πράγματα στο άμεσο μέλλον. Κάποια θα μείνουν στην Ευρωζώνη, κάποια θα μείνουν εκτός. Και χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειαζόμαστε να δουλεύει και να εργάζεται για να λειτουργεί για όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για την Ευρωζώνη. θα δημιουργηθούν πολλά περισσότερα προβλήματα αν, έχει μεγαλύτερη επιρροή, αν έχουν μεγαλύτερη επιρροή οι χώρες της Ευρωζώνης. Σας παρακαλώ λοιπόν να διαβάσετε τις τροπολογίες μου για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, για τη συμμετοχή και για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι λειτουργική για όλα τα κράτη-μέλη. Μελετήστε προσεκτικά λοιπόν τις προτάσεις μου και προσπαθήστε να δώσετε μία λύση, γιατί πραγματικά χρειάζεται να δώσουμε μία λύση στο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ashley Fox. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ashley Fox. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Δεν θα μάθετε, δεν θα εκπλαγείτε αν μάθετε ότι διαφωνώ αρκετά με την έκθεση αυτή, για να μην πω κάθετα. Δεν θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει κυβέρνηση της Ένωσης και δεν θέλω πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια. Ούτε τώρα ούτε τα ήθελα όταν τα είχε προτείνει ο Άντριου Ντάφο να ήταν βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ όμω με την παράγραφο 39 όπου λέμε να έχει μία έδρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι δύο. Σε αυτό συμφωνώ. Το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δύο έδρε και πηγαίνω έρχεται μεταξύ των δύο, σπαταλώντα χρόνο, χρήμα και εξοδεύοντα διοξίδιο του άνθρακα, το μόνο που κάνει είναι να καταφέρνει πλήγμα κέραιος στη φήμη αυτού του θεσμικού οργάνου. Έχουμε την έκθεση Fox Hafner. Το 2012 εγκρίθηκε και ε, θέλουμε συνταγματική αλλαγή έτσι ώστε να είναι μία μόνο έδρα και αν υπάρξει τέτοια απόφαση, η συνταγματική αλλαγή είναι να μπορεί να το αποφασίσει το ίδιο το Κοινοβούλιο. Δηλαδή Υπήρξε έτοιμα να υπάρξει έκθεση που θα προτείνει αλλαγή των συνθηκών και η διάσκεψη των Προέδρων δεν έδωσε το πράσινο φως, γιατί υποτίθεται ότι το θέμα αυτό θα το κάλυπτε η έκθεση Φερχόφστατ. Και δυστυχώς Γκί δεν το κάλυψε στο θέμα. Επανέλαβε στη θέση, δεν πρότεινε αλλαγή των συνθηκών, κάτι το οποίο ψήφισε το Κοινοβούλιο το 2012 και κάτι το οποίο η δική μας Επιτροπή ζήτησε να τεθεί επιτάπητο στην αρχή της κοινοβουλευτική θητείας. Ξέρετε, αν ρωτήσετε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα δείτε ότι η ισχυρή πλειοψηφία εξ αυτών θέλει μία και μόνη έδρα και να αποφασίσει το Κοινοβούλιο ποια θα είναι αυτή. Κάθε φορά που πάει όμως το θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων, εκεί ε, χαλάει λίγο η συνταγή, να μην ενοχλήσουμε τους Γάλλους, να μην τους ταράξουμε και τελικά δεν συζητείται ποτέ το θέμα από τη διάσκεψη των Προέδρων. Συμφωνείτε λοιπόν με το 39, αλλά δεν του δίνετε συνέχεια. Νομίζω ότι η λύση είναι αρκετά απλή και καλούνται να αναλάβουν δράσεις οι συντονιστές. Να επαναλάβετε το αίτημά σας στη διάσκεψη των Προέδρων να πυροδοτηθεί η έναρξη αυτής της ε, αλλαγής των ζηθικών. Μπορεί το Κοινοβούλιο να, μας να το κάνει, να το θέσει επιτάπητος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μία πρόταση αλλαγή τη συνθήκη, την οποία θα πρέπει να εξετάζει το Συμβούλιο και να τους προκαλέσετε να την καταψηφίσουν. Γιατί ιδελιώ θα είναι πάντοτε δύσκολο και πάντοτε θα βρίσκονται κάποιοι που δεν θα θέλουν να, να ταράξουν τους γάλους Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Να μην σας θυμίσω πόσες φορές έχουμε παγώσει το έργο μας για να μην ταράξουμε τους Βρετανούς. Ε, σε αυτό έχουμε παράδοση, ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί ήρθε η ώρα, θέλετε κάτι να πείτε, παρακαλώ. Ναι. Να αντιδράσω σε διάφορα τηρήσεις που έγιναν. Και να επαναλάβω όμως ότι την επόμενη εβδομάδα θα προτείνω διάφορες συμβαστικές τροπολογίες που θα βασίζονται στις τροπολογίες που έχω λάβει και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε με τους κοιόδης εισηγητές να συνεργαστούμε μετά και να κάνουμε πολύ έντονες επαφές την επόμενη εβδομάδα για να φτάσουμε σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Να επαναλάβω ότι στην έκθεση ε, εμπνεύστηκα από τους θεμελιώδεις πατέρες, από τους ιδρυτικούς πατέρες αν έχετε πρόβλημα με τον Αλτιέρο Σπινέλη, τον Μπόλαν Ρισπακ και τον κύριο Βραντάνο, ε, τι να σας πω. Αυτοί στη δεκαετία του 50, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ας πούμε, έκαναν την, μίλησαν για την ΕΟΚ, για την Αμυντική Ένωση κτλ. Δεν συζήτησαν μεταξύ τους τι είδους πολιτικές ε, θα πρέπει να προωθήσει η Ένωση. Είπαν, ο ένας ήταν σοσιαλιστής, ο άλλος ήταν κομμουνιστής και ο άλλος ήταν κομμουνιστής. Μόνο οι φιλελεύθεροι απουσίαζαν τότε από το κλαμπ. Ναι, ναι, έτσι ήταν Mercedes. Δεν άρχισαν να λένε χρειαζόμαστε λίγο από αυτό, χρειαζόμαστε λίγο από εκείνο, χρειαζόμαστε περισσότερη λιγότερη ε, λιτότητα, περισσότερο και ενσιασμό, ε, και ε, όχι. Είπαν θέλουμε μία ένωση. Οικονομική, αμυντική και πολιτική ένωση. Και χρειαζόμαστε και ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 53, όχι το 79. Όλα είχαν προβλεφθεί τότε. Δεν ξέρω αν η γραμματεία της Επιτροπής ΑΦΚΟ μπορεί να στείλει σε όλα τα μέλη της ΑΦΚΟ το πρώτο σύνταγμα της ε, Ευρώπης που εγκρίθηκε με ομοφωνία και πέντε αποχές από όλα τα μέλη της ad hoc συνέλευσης που εκπροσωπούσαν τα έξι ιδρυτικά κράτη της Επιτροπής Άνθρακα και Χάλιβα. Διαβάστε το, είναι θαυμάσιο ανάγνωσμα. Για να αναρωτηθείτε τι το θαυμάσιο έγινε το τεστικέ του 50 και που εμείς δεν έχουμε μπορούμε να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία κατά της, ε, για την ε, Τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε μία αμυντική ένωση, γιατί να μιλάμε για αυτήν και λοιπά και λοιπά. Το λέω γιατί άκουσα παρατηρήσεις ότι δεν μιλάς για το περιεχόμενο των πολιτικών. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Δεν είναι ο σκοπό αυτή τη έκθεση να μιλήσω για τι πολιτικέ και το περιεχόμενό του. Όπω δεν ήταν ο σκοπό του Σπινέλη, του Σπακ, του Μπραντάνο και όλων των υπολείπων να αρχίσουν μια συζήτηση μεταξύ του για τι πολιτικέ τη Ένωση. Όχι. Μιλούσαν για το θεσμικό πλαίσιο. Όταν έχει ένα καλό θεσμικό πλαίσιο, όταν το στήσει, τότε αρχίζει να πτήσει τι πολιτικέ σου. Αν οι χριστιανοδημοκράτε, οι φιλελεύθεροι ας πούμε ε, έρθουν στην εξουσία θα είναι διαφορετικό από το αν έρθουν οι, οι σοσιαλιστές κτλ. Πάντως αυτό είναι το θέμα. Θέλουμε το θεσμικό πλαίσιο. Γι' αυτό μιλάμε. Γιατί μιλάμε για το θεσμικό μέλλον της Ένωσης. ένα τέτοιο πλαίσιο που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που μας ταλανίζουν. Γιατί, ας τα πούμε ξεκάθαρα, γιατί φτιάξαμε την ε, έκθεσή μου, την έκθεση Μπρέσο Μπροκ, γιατί έχουμε διάφορες προκλήσεις και δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις αντιμετωπίσουμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το καθάρισμα των τραπεζών στην ε, Ευρώπη. Πού έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα πρόβλημα με τράπεζες οι οποίες δεν είναι εξυγιασμένες. Ενώ στη ΣΥΠΑ, ήδη το 2014, οι ΗΠΑ έβαλαν λεφτά και συνεχεία αυτά τα λεφτά δόθηκαν πίσω στους ε, φορολογούμενους, ενώ εμείς ακόμα δεν έχουμε καθαρίσει τράπεζες. Το πρόβλημα δεν έχει λήξει. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε τεράστια χρηματοπιστωτικά προβλήματα στην Ένωση, λόγω του γεγονότος ότι οι τράπεζες μας έχουν ε, πρόβλημα. Γιατί, γιατί δεν είχαμε από την αρχή την Τραπεζική Ένωση. Και ακόμα και σήμερα δεν είναι πλήρης η Τραπεζική Ένωση. Και δεν έχουμε και ένα ταμείο για να παρέμβει σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα με κάποια τράπεζα στην ε, Ευρώπη. Επομένως, το θεσμικό μας πλαίσιο δεν είναι σωστό το θεσμικό πλαίσιο που χρειαζόμαστε. Δεύτερη παρατήρηση. Ας μην ξεγελιόμαστε. Υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι μιλάτε ότι προωθείται μια υπερβολική συγκεντρωτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μιλάτε για συγκεντρωτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι το 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Διάφοροι λένε υπερσυγκέντρωση ας πούμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέμβαση στα πάντα. Με το 1% του προπολογισμού, ας πούμε, με το 1% του ΑΕΠ, του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Το 80% αυτό του 1% πηγαίνει πίσω στα κράτη-μέλη. Οι συνεισφορές των κρατών μελών επιστρέφουν πίσω. Και από το 20% που μένει, το 0,2% δηλαδή του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, το 0,06% το χρειαζόμαστε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για τους υπαλλήλους, για τις, ε, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς κτλ. Δηλαδή, τελικά τα λεφτά που έχουμε στη διάθεσή μας για να, φτιά, για να προωθήσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα και project ας πούμε, είναι το 0,14%. Σταματήστε λοιπόν αυτό το, αυτό το τροπάρι. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπλοκάρει τα πάντα, που παρεμβαίνει στα πάντα, που χρηματοδοτεί τα πάντα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτά τα λένε οι ευρωσκεπτικιστέ. Και τελικά και οι φιλοευρωπαίοι πιστεύουν ότι είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό είναι το πρόβλημα τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι τελικά κυριαρχεί ο ευρωσκεπτικισμός. Και ακόμα και αυτοί που είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετούν αυτά τα επιχειρήματα. Τώρα, για πιο συγκεκριμένε παρατηρήσει που ακούστηκαν. Μίλησα για αυτό το καθεστώ συνδεδεμένου κράτου. Ε, για, το, το έκανα για να έχουμε ένα πλαίσιο για να βάλουμε ας πούμε μέσα εκεί τις ε, εταιρικέ σχέσεις. Φυσικά άλλη σχέση θα έχουμε με την Τουρκία, άλλη με την Ουκρανία, άλλη με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει ποια θα είναι αυτή η εταιρική σχέση με, την, με το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να δούμε καταρχά την πρόταση τη Βρετανική κυβέρνηση. Αλλά τουλάχιστον είναι απαραίτητο να πούμε ότι είναι από τη μία τα μέλη και από την άλλη τα συνδεδεμένα κράτη. Ότι υπάρχουν διαφορετικέ εταιρικέ σχέσει με διαφορετικέ χώρε, προφανώ συμφωνώ, αλλά υπάρχουν ελάχιστε προποθέσει που θα πρέπει να τι σέβονται όλοι αυτοί οι εταίροι. Αυτή είναι η ιδέα και θα κάνω μια πρόταση για να ορίσω αυτή την, ε, τις ελάχιστες ας πούμε, προϋποθέσεις και συνθήκες. Τώρα, το τι είναι μέλος, ποιος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αν θες να συνεχίσεις τον πολλαπλασιασμό, opt-in, opt-out, ε, μέσων συνεργασίας κτλ, εμπρός. Κάντε το. Αλλά εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα δεν χρησιμοποιούμε τα συστήματα. Γιατί? Εγώ θυμάμαι τις διαπραγματεύσεις για την Ίκαια. Για να διευκολύνουμε, ας πούμε, την ενισχυμένη συνεργασία, τη διαρθρωμένη συνεργασία. Επίσης πάλι, ας πούμε, στη συνθήκη της Λισαβόνας απαλύναμε τις προϋποθέσεις. Στην πραγματικότητα, όταν έχουμε προβλήματα, τα Όπω α πούμε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, τα ξεπετάγουμε, τα, λύνουμε εκτό τη συνθήκη. Αυτό γίνεται. Και οι αρνητικέ συνέπειε είναι ότι δεν υπάρχει ο συνήθι και δεν εφαρμόζεται ο συνήθι και απαιτούμενο δημοκρατικό έλεγχο. Και γι' αυτό θα πρέπει να βάλουμε στην έκθεση Μπροκ Μπρέσο ένα κατάλογο από συνεργασίες και πολιτικές που θα θέλαμε να επανεισάγουμε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτή είναι η πραγματικότητα η σημερινή. Δεν θέλω να σας κουράσω με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι. Εάν τον δείτε συνολικά, θα δείτε πόσα λεφτά είναι εκτός του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτά που είναι εντός. Σε... Στην έκθεση που θα δημοσιευτεί μέχρι το τέλος του 2016, είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της, θα έχουμε μία απεικόνηση του πώς μοιάζει ο ευρωπαϊκός προπολογισμό είναι πολύ χειρότερος από τη διαφάνεια που μου έδειξε ο κ. Κόρμπετ πριν από λίγο για τα διάφορα, διάφορα opt-in, opt-out, ε, ενσχημένες συνεργασίες, κύκλους, παρακυκλάκια, ομόκεντρους κτλ. που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πλουστεύσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ότι αύριο όλοι θα υιοθετήσουν το ευρώ. Και ούτε το εννοούμε κάτι τέτοιο και ούτε το θέλουμε. Απλώς τουλάχιστον να υπάρχει μια κατεύθυνση και να λένε ότι η κανονική, η συνήθι κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι κάθε κρατό μέλο συμμετέχει σε όλε τι πολιτικέ τη Ένωση. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Και εμεί θεωρούμε ότι το φυσιολογικό είναι το αντίθετο. Γιατί δημιουργήσαμε τόσα πολλά opt-in και out παραδείγματο στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι θα κάνουμε στο επόμενο. Θα πρέπει να ξεφορτωθούμε, ας πούμε, την ε, μείωση, το rebate, το βρετανικό. Ή θα, θα... θα συνεχίσουμε, ας πούμε, να εφαρμόσουμε την ε, μείωση, με επιστροφή δηλαδή, που δίναμε στη Βρετανία, όταν φύγει η Βρετανία. Εάν δεν έχουμε αυτή τη μείωση, η επιστροφή, ας πούμε, δεν, δεν μπορούμε να έχουμε επιστροφή στην επιστροφή. Ίσως βρείτε μια άλλη λύση. για τις οικονομικές ανάγκες ή για τις επιθυμίες μας. Αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργούμε επιστροφές επί επιστροφών, επί επιστροφών κτλ. Θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των εξαιρέσεων. Ας συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί αλλιώς θα γίνει μια έκρηξη εξαιρέσεων, ένας πολλαπλασιασμός εξαιρέσεων και στον προπολογισμό και αλλού. Για τη ρήτρα σύγκληση. Συμφωνώ. Θα δούμε με τους σκιώδες εισηγητέ ε, πώ θα τα βρούμε, αλλά εγώ δεν μιλούσα μόνο για την οικονομική και χρηματοπιστωτική διάσταση, αλλά και για τα αθρολογικά θέματα και για τα κοινωνικά θέματα και για τα συνταξιδοτικά θέματα. Σύγκληση. Η ιδέα είναι να έχουμε μια τέτοια σύγκληση. Αυτό το είχαμε υιοθετήσει την ιδέα της σύγκλησης σε διάφορα ψηφίσματα εδώ στο Κοινοβούλιο που συμφωνήσαμε τα τελευταία χρόνια. Um, uh, Από εκεί και πέρα. Για την πράσινη, την κόκκινη και την πορτοκαλί κάρτα πρέπει αυτά να τα συζητήσουμε περισσότερο σε βάθος. Με τους διάφορους και όδες εισηγητές σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρώσω με κάτι που αναφέρθηκε στην τελευταία παράγραφο για τη συνέλευση. Και συνέλευση να μην έχουμε, να έχουμε έναν σε βάθος προβληματισμό τουλάχιστον. Θα υπάρξει μια διαδρα... διαδρομή διαπραγμάτευσης με τους Βρετανούς. Να ανοίξουμε ένα δεύτερο διάδρομο προβληματισμού για τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω ότι πρέπει αύριο να συγκληθεί συνέλευση αλλά ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις για το Brexit να ξεκινήσει ένας προβληματισμός έτσι ώστε στο τέλος αυτής της διαδικασίας και όταν θα υπάρξει συμφωνία με τη, Μεγάλη Βρετανία να έχουμε μια σαφή ιδέα για το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν θα δώσω ε, το λόγο σε κανέναν, ζητώ συγγνώμη, γιατί έχουμε μόνο πέντε λεπτά για την έκθεση Μπροκ. Ας σας δώσω το λόγο. Από ό,τι καταλαβαίνω θα συναντηθείτε με τους σκιώδεις εισηγητές για να ψηφίσουμε στις 21. Λοιπόν, προχωρούμε τάχιστα. Έλμαρ, παρακαλώ ε, και τους λοιπούς, ε, μπορείτε να μιλήσετε το συντομότερο δυνατό και το λιγότερο δυνατό όταν πάρετε το λόγο. Έχουμε πέντε λεπτά μόνο. Ησυχία παρακαλώ. Μια στιγμούλα. Dunque, ε, noi abbiamo inviato a tutti... Στείλαμε σε όλους τους κοιόδης εισηγητές μια πρόταση πολύ μακροσκελή, πολύ περίπλοκη, περίπλοκη με συμβιβασμούς για το σύνολο των τροπολογιών που υποβλήθηκαν. Προφανώς ε, μιλάω για τις τροπολογίες που σέβονται τη λογική της έκθεσής, της μας. Μία έκθεση που είναι φιλοευρωπαϊκή, που θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία σας και αγράφησε ο, ο Φερχόφσταντ τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, στο εσωτερικό των ε, υπαρχουσών συνθήκων ή με τροποποίηση ή με νέα συνθήκη σε κάποιο βαθμό. Λοιπόν, πού έχουμε φτάσει. Χτες είχαμε κάποιες δυσκολίες στις συζητήσεις για τις τροπολογίες. Ζητήσαμε από όλου τους συναδέλφους, τους κοιόδης εισηγητές δηλαδή, να μας πούν γραπτός τι αλλαγές θέλουν να επιφέρουμε μέσω συμβαστικών τροπολογιών και να μας πούν να συμφωνούν ή διαφωνούν ε, με τις προτάσεις που υποβάλαμε. Λάβαμε λοιπόν μια σειρά από παρατηρήσεις που θα μας οδηγήσουν σε κάποιες αλλαγές. Όταν συμφωνήσουμε. Θα μας οδηγήσουν δηλαδή σε συμβαστικές τροπολογίες. Και ελπίζω μέχρι αύριο να στείλουμε τις συμβαστικές τροπολογίες σε όλους τους σκιώδες εισηγητές. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι σκιώδες εισηγητές που δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Εάν μου το ζητήσουν όμως κάποιοι άλλοι σκιώδες εισηγητές να συζητήσουμε κάποια θέματα, θα, θα τα συζητήσουμε. Εάν όμως ε, δεν μου ζητηθεί κάτι τέτοιο, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Έλμαρ, θες να προσθέσεις κάτι ή σε κάλυψε η Mercedes. Οι σκιώδεις ηγητές θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Το βασικό είναι να φτάσουμε στους καλύτερους δυνατούς συμβασμους Αυτή η δουλειά θα γίνει με συνεννόηση μεταξύ των ομάδων. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να ψηφιστεί 21 Νοεμβρίου, αργά με στην ημέρα. Πάμε τώρα στην, στο τελευταίο σημείο. Ο, συγγνώμη, ο Έλμαρ, παρακαλώ. möchte dann doch noch klarstellen, wie gesagt, es geht morgen früh raus, äh, Vorschläge auf unsere ursprüngliche... Ναι. Θα ξαναδούμε τι προτάσει και είναι πολύ καλά τα σχόλια που έχουμε πάρει Μέχρι αύριο το βράδυ μπορεί κανείς να κάνει και άλλες ε, προτάσεις. Αν το κάνουμε έτσι ε, με δύο γύρους, τότε δεν θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε καινούριες τροπολογίες την επόμενη εβδομάδα. Δεν μιλάμε για την ε, θέση σε ισχύ νέων χρονικών περιόδων και προθεσμιών για υποβολή τροπολογιών. Καλώς. Συμβιβαστική λύση μέχρι ε, αύριο προς το τέλος της ημέρας μπορεί να υπάρξει. Μόνο αυτό. Δηλαδή έχετε ε, χρόνο μέχρι αύριο βράδυ να στείλετε ιδέες για τις συμβαστικές τροπολογίες. Όχι όμως καινούργια θέματα, δεν μπορούν να ανοίξουν για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η εξέταση αυτού του σημείου της μερίσιας διάταξης.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 Καταληκτική, καταληκτική προθεσμία για την έκθεση Ραμό Χαουρέγγι ήταν σήμερα για να υποβάλλετε τροπολογίες, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα το σύστημα, άρα δίνουμε παράταση μέχρι αύριο στις 6 το απόγευμα. Έκθεση Ραμόν Χαουρέγγι. Ευχαριστώ. Ας προσπαθήσω να ανοίξω το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε τον Άντριου Νταφ και τον Μάικλ Έμερσον. Συνεχίζεται η Βρετανική σάγκα, ο Βρετανικός μύθος. Οι αβεβαιότητες αντικαθίστανται με, από νέες αβεβαιότητες. Κάποια στιγμή θα υπάρξει κόπωση από το Brexit. Έχουμε ορίσει κάποιους αρμοδίους ως κοινοβούλιο, αλλά όλα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ε, δεν έχουμε προβληματιστεί ε, επαρκώς πιστεύω. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να έχουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως εξηγούσα λοιπόν στο Μάικλ και στον Άντριο, στόχος μας είναι και σχέδιο μας είναι να συνεχιστούν οι συζητήσεις, να προσπαθήσουμε να λύνουμε τα προβλήματα όπως θα προκύπτουν και να κομίσουμε νέα γνώση, νέες ιδέες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δικές σας ιδέες, Μάικλ και Άντριου, εντάσσονται σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτή την προσπάθεια. Ε, γι' αυτό σας έχουμε εδώ για να εμπλουτίσετε τον προβληματισμό μας. Ποιος θα μιλήσει πρώτος, ο Άντριου. Καλώς. Έχετε το λόγο. Το λόγο ε, θα έχει ο Άντριου Ντάφ, τον οποίο φυσικά δεν χρειάζεται να σας παρουσιάσω. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα το ότι βρίσκομαι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων που είναι και η πιο σημαντική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο λόγος για τον οποίο είμαστε εμείς εδώ απόψε είναι εξαιρετικά θλιβερός και θα έλεγα καταστροφικός για το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά τα συμβάντα και τις ε, αντικσοότητες, τις αμφιλεγόμενες απόψεις, τις διαμάχες που έχουν προκύψει σε βάθος χρόνου, είναι απαραίτητο το Κοινοβούλιο να έχει συνολική συνεκτική προσέγγιση σε αυτό το οποίο ήδη αποκαλείται η σάγκα του Brexit. Έχω καθίσει στα έδρανα που κάθονται αυτή τη στιγμή ο κύριος Φερχόφστατ και ο κύριος Μπρόκ. Όπως γνωρίζετε. Και έχω γράψει και μια έκθεση. Brexit ή Brexit, άνω κάτω τελεία, τι μέλη γενέστε, τι έπεται. Είναι κάπως μακροσκελής η αναφορά μου αυτή, αλλά είναι μακροσκελής και εκτείνεται σε πολλές σελίδε, ε, ακριβώς γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά περίπλοκο και λεπτό. Ξέρετε, στο Λονδίνο λέγεται ότι το Brexit σημαίνει Brexit. Ενώ εδώ, στις Βρυξέλλες, λέγεται ότι μπορεί να υπάρξουν μη συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για όσο καιρό εκρεμεί η το αίτημα για τη θέση σε ισχύ και εφαρμογή του άρθρου 50 των συνθηκών. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι δημιουργείται ένα νομικό κενό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε παραλυσία. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, προσπαθώντας να γεφυρώσει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα, το οποίο βαίνει αυξανόμενο. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα έλεγα ότι θα πρέπει το Βρετανικό Κοινοβούλιο να διευκρινίσει κάποιες από τις επιλογές που θα μπορούσαν να ήταν αποδεκτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καθορίσει ποιες από, α, επιλογές είναι αποδεκτές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες θα μπορούσαν να είναι να είναι ε, αποδεκτές. Έχουμε την επιλογή της Νορβηγίας ή του Καναδά ή της Τουρκίας, δηλαδή οι συμφωνίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αντίστοιχες χώρες. Όμως, αυτό δεν οδηγεί σε τίποτα το ρεαλιστικό, τίποτα το επικοδομητικό και τίποτα το δημιουργικό. Ενώ εμεί χρειαζόμαστε και τα τρία αυτά προκειμένου να υπάρξει μια οριστική διευθέτηση της ε, προβληματικής αυτής σχέσης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, το Κοινοβούλιο οφείλει να καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, να μιλήσει με μεγαλύτερη ευγλωτία, με μεγαλύτερη αμεσότητα, πολύ μεγαλύτερη από όσο μπορεί να το πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Και θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρατε κάτι τέτοιο. Μιλούσε δηλαδή με την παρησία που λείπει από τα άλλα θεσμικά όργανα. Και πιστεύω ότι Πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια συνεκτική θέση για το ποιες θα είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ηνωμένο Βασίλειο σε βάθος χρόνου. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρξουν προτάσεις από τις Βρυξέλλες. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν αποφάσεις στην ομολογία του δικαστηρίου και τις περιγράφω στην έκθεση που σας έχω διαβιβάσει. Όλα αυτά συντείνουν στην δημιουργία σύγχυσης και περαιτέρω καθυστερήσεων. Και το πρωταρχικό ζήτημα έχει να κάνει με το προνόμιο της κυβέρνησης, την και ε, νομή της εξουσίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης. Είναι εγχώριο το ζήτημα των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο και ε, δεν θα πρέπει να εμπλακεί στις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, το αποτέλεσμα αυτών των αντιφάσεων μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η απόφαση αυτή του δικαστηρίου, του σχετικού, του Βρετανικού, η οποία έχει και άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της διαπραγματευτικής διαδικασίας του Brexit και στη χρονική συγκυρία κατά την οποία αυτό συμβαίνει. Αυτή ε, ε, πυροδοτείται και λαμβάνει χώρα. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι το εξής. Ε, τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο το άρθρο 50 και η κοινοποίηση για τη θέση σε ισχύ του άρθρου 50 μπορεί να αποσυρθεί. από το Ηνωμένο Βασίλειο και αν θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή άποψης. στο Βρετανικό Δικαστήριο και η ενάγουσα αρχή και το, η κυβέρνηση συμφώνησαν ότι δεν είναι θέση αυτή, ε, ότι δεν είναι δηλαδή μετακλητή η απόφαση. Θα πρέπει να ζητηθεί η θέση σε ισχύ του άρθρου 50, είτε αυτή καταλήξει σε συμφωνία, είτε καταλήξει σε μη συμφωνία. Και αν καταλήξει σε μη συμφωνία, τότε οι συνθήκες απλά θα σταματήσουν να ισχύουν. Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η απόφαση και αυτό δέχθηκαν και τα δύο διάδικα μέρη. Εγώ όμως και πολλοί άλλοι δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η ορθή νομική ερμηνεία του άρθρου 50 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως σε δεύτερο βαθμό στο ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου όταν κριθεί αυτή η υπόθεση να ε, προκύψει και να ανακύψει αυτό το ζήτημα. Και αν υπάρξει επίκληση και αναφορά σε αυτό το ζήτημα τότε αναπόφευκτα θα γίνει και αναφορά στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν θα γίνει προαιρετικά, είναι, υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτικό αυτό. Και αν τούτο συμβεί, τότε και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα μπορούσαν να ε, παρέμβουν στη δίκη να ε, δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής και να ε, προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τη διαδικασία μέσω της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να ζητήσει την ανάκληση της θέσης σε ισχύ και σε εφαρμογή του άρθρου 50. και θα μπορούσαν να υπάρξουν οι συνθήκες για θετική έκβαση από πλευρά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι να πάψει η διαδικασία του Brexit. Το ηρωνικό είναι ότι παρά την έκβαση της διαδικασίας στο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει το ε, Βρετανικό Κοινοβούλιο να αποφασίσει να θέσει σε ισχύ το άρθρο 50. Δεν υπάρχει βεβαιότητα επ' αυτού. Είναι μεγάλη η πλειοψηφία και στη Βουλή των Κοινοτήτων και στη Βουλή των Λόρδων. Ότι δηλαδή το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος οφείλει να ε, εφαρμοστεί, να λάβει χώρα. Είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουμε εδώ στην Ευρώπη να ε, μιλάμε ε, το, για το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Βασίλειο θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ίσως φύγει. δεν είναι... δεν είναι θα μπορούσε να φύγει, είναι ότι θα φύγει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση όμως οι πολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραστικά και μπορούν να αλλάξουν έτσι περαιτέρω στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι ε, μπορεί να υπάρξει αλλαγή στάσης και πλεύσης. Σε κάθε περίπτωση το άρθρο 50 ε, θα τεθεί σε ισχύ, θα ζητηθεί δηλαδή η θέση σε ισχύ και σε εφαρμογή του άρθρου 50 και στο τέλος της επιτυχημένης της περίοδου διαπραγμάτευσης μετά από δύο χρόνια μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία και θα χρειαστεί αυτή η συμφωνία τη στήριξη και την επικύρωση, αν θέλετε, από το Κοινοβούλιο το Βρετανικό. Πρέπει να τονίζω συνεχώς το, γεγο... το εξής γεγονός. Η συμφωνία αυτή καθεαυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με τα τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να διευκρινιστούν έτσι ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να απεμπλακεί από τα δικαιώματα και από τις υποχρεώσεις του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω συνοψίσει τα άρθρα στην παράγραφο 2,3 στο έγγραφό μου. Κάποια ζητήματα είναι περίπλοκα, έτσι όπως θα αναφέρω στο εδάφιο 2,3 της έκθεσής μου και κάποια άλλα είναι πολύ πιο απλά. Θα πρέπει να υπάρξει μερική συμφωνία για αυτό το οποίο το άρθρο περιγράφει ως το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων. Και η πρόταση που διατυπώνω, όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι, είναι η εξής. Αυτή η επιμέρους συμφωνία να διατυπωθεί και να συμπεριληφθεί σε ορισμένα συμπεράσματα ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. και όχι ως επίσημο μέρος ε, βάση του άρθρου 50. Γιατί εάν στη συμφωνία βάση του άρθρου 50 συμπεριλάβουμε ουσιαστική έκφραση και περιγραφή ε, της τελικής ρύθμισης και της τελικής διευθέτησης ελοχεύει ο κίνδυνος το άρθρο 50 να ερμηνευθεί ως μεικτή συμφωνία και άρα να απαιτήσει την ομοφωνία από όλα τα κράτη-μέλη και την έγκριση από όλα τα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου να ισχύσει. Ακόμα και μέσω δημοψήφισμάτων και είχαμε και ένα, πολλή εμπειρία γι' αυτό. Γι' αυτό και προτείνω λοιπόν τα τεχνικά να μπουν σε συμπεράσματα του Συμβουλίου και όχι στη συμφωνία που θα επικαλείται το άρθρο 50. Γιατί ε, αλλιώς θα πρέπει να περάσει από τα εθνικά κοινοβούλια με δημοψηφίσματα και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι αυτό σημαίνει. Τα συμπεράσματα θα πρέπει να διατυπωθούν ως απόφαση του Συμβουλίου και εκεί χρειάζεται η ε, ειδική πλειοψηφία, απλά. Απλή ειδική πλειοψηφία και δεν χρειάζονται έγκριση από 27 κοινοβούλια ή 27 δημοψηφίσματα προκειμένου να ισχύουν. Θα πρέπει αυτό να το γνωρίζουμε, να το έχουμε συνειδητοποιήσει και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία συμφωνία όσο δυνατόν πιο καθαρή και πιο απλή μπορούμε. Φυσικά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα σύστημα για την προσωρινή μεταβατική περίοδο από την φάση στην οποία βρισκόμαστε δηλαδή τώρα μέχρι το Brexit. μέχρι την τελική, δηλαδή το τελικό Brexit. Θα είναι οι ρήτρε διάδρομοι. Ορισμένες μπορεί να έχουν χρονικό περιορισμό, αλλά ο βασικός στόχος αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας, που θα είναι πολύ δύσκολο να διαμορφωθεί, θα είναι να μεταβούμε τελικά όλοι μας το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ένωση των 27 στο σημείο που θέλουμε να πάμε. Στο σημείο που θα συμφωνήσουμε ότι θέλουμε να πάμε. Μειώνοντας τις παράπλευρες απώλειες. που θα προκύψουν εάν πέσουμε στον κρεμό όλοι Εγώ και ο Μάικλ Έμερσον συμφωνούμε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε ένα υπόδειγμα, ένα μόρφωμα και το προηγούμενο είναι η συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία. Δεν μιλάμε για ένα καθεστώς συνδεδεμένου κράτους, όπως αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως με την έκθεση Φερχόφστατ. Είναι μία πρακτική και πλήρης λύση σε ένα πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν πολλές απλές λύσεις. Έχουμε ένα προηγούμενο, συμφώνησε η Ουκρανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε μια τέτοια συμφωνία το 1954 με την παλιά κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Άρα μπορεί να γίνει. και ο Μάικλ θα σας εξηγήσει πιο αναλυτικά και θα σας περιγράψει τη μορφή που έχουμε στο μυαλό μας. Ο Μάικλ Έμερσον που είναι ερευνητής έχει το λόγο. Χαιρόμαστε που ξαναέρχεσαι εδώ στο Κοινοβούλιο Μάικλ. Ευχαριστώ Ντανούτα. Όπως είπε και ο Άντριου, θα μιλήσω για το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου που θα διέπει τις μελλοντικές σχέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε ένα άδειο ποτήρι. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πει πολλά, λίγα έχει να λέει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα πει τίποτα μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο να πάρει θέση να παίξει την πρώτη μπαλιά. Η Πρωθυπουργό είπε, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ε, ε, να αποκλείσουμε διάφορα πράγματα. Θέλουμε το καταλληλότερο μοντέλο το οποίο είναι καλύτερο για την ε, Βρετανία. Πολιτική ρητορία είναι αυτή. Η συζήτηση για τα μοντέλα είναι πολύ αποτελεσματική όταν εντοπίζουμε τα μοντέλα, όταν τα ξέρουμε αυτά τα μοντέλα. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να συζητήσουμε την ουσία των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων χωρίς να πνιγούμε με λεπτομέρειε. Υπάρχουν πέντε γνωστά μοντέλα που κυκλοφορούν και κάθε ένα από αυτά έχει σημαντικά μειονεκτήματα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και το έκτο, το οποίο ανέφερε ο Άντριου, θα στο συζητήσω. Λοιπόν, για τα πέντε πρώτα. Η απλή συμμετοχή τύπου ΠΟΕ, αλλά αυτό σημαίνει βλάβη στην πρόσβαση και προβλήματα στην πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στην ε, νέα αγορά. Ε, το καθεστώς ε, EA είναι ασύμβατο για τον έλεγχο της μετανάστευσης. το σουηδικό μοντέλο δεν θα είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ακανδικό μοντέλο θεωρώ ότι είναι άσχετο γιατί αγνοεί τεράστια κομμάτια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Καθώς βέβαια και η Τελωνιακή Ένωση που περιορίζει τις δυνατότητες. Λοιπόν, έχουμε και το έκτο μοντέλο, αυτή την ε, συμφωνία ανάλογη με της Ουκρανίας. Το θέμα δεν είναι η ιστορία με την Ουκρανία, το θέμα είναι πώς θα διαμορφώσουμε ή μάλλον το θέμα είναι η δομή του ευρωπαϊκού δικαίου που μπορεί να μην ε, εφαρμόζεται και να μην ισχύει στο τρίτο μέρος. Τα χαρακτηριστικά τα οποία ενδιαφέρουν το, τη Βρετανία είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Επίσης, ε, για τρεις από τι ελευθερίε ελευθερίες της διαπραγματεύσεις είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά όχι για, τα, για τους εργαζόμενους. Και έχει επίσης και νομικά και θεσμικά στοιχεία που μπορεί να είναι σημαντικά. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συζητάει τις ε, εναλλακτικέ μυστικά. Στο μεταξύ ε, γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα. Ε, η υπόθεση Νισάν είναι η πιο σημαντική, καθώς και η απόφαση του του Δικαστηρίου για το άρθρο 50, που αποκαλύπτει ότι μια πλειοψηφία των βουλευτών θα θέλανε ένα ήπιο μοντέλο Brexit για την επιστολή ενεργοποίησης του άρθρου 50. Ο κύριος Κάρλο Ντόνζον έφυγε από το, την πρωθυπουργική κατοικία λέγοντας ότι οποιαδήποτε και, θα είναι, και αν είναι το αποτέλεσμα, η δική του εταιρεία δεν θα έχει πρόβλημα. Οι λεπτομέρειε δεν είναι γνωστέ. αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε αν όλες αυτές οι διαβαβαιώσεις έχουν και νομική ισχύ. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την έχουμε συμβουλευτεί για αυτό το θέμα. Τώρα, μήπως αυτό θα πιέσει την κυβέρνηση να πει λίγο περισσότερα. Ο Υπουργό για τον Brexit είπε θέλει ε, να μην υπάρξουν γραφειοκρατικά εμπόδια και φυσικά μηδενικούς δασμούς στο Brexit. Αυτό τι σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει τελωνιακή ένωση, μπορεί να σημαίνει ε, απλά, ε, ε, DCFTA τύπου Ουκρανίας ή μπορεί να σημαίνει επίσης ένα συνδυασμός και τελωνιακή Ένωσης και ε, δελεχούς ε, ζώνης ελευθέρου εμπορίου. Για το περιεχόμενο τώρα. Είναι πολύ ουσιαστικό. Έχουμε δύο συμφωνίες ε, σύνδεσης. Μία είναι DCFTA και άλλη, το άλλο τύπος είναι οικονομική συνεργασία. Το DCFTA έχει 10 κεφάλαια τουλάχιστον, τα οποία είναι γνωστά σε όλους σας αλλά μπορούν να εντοπιστούν ως ελάχιστες προϋποθέσεις που μπορεί να περιμένει ο καθένας ε, να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ελληνικούς δασμούς, ε, τελωνιακές διαδικασίες, τεχνικά πρότυπα για τα αγαθά, κανόνες αντι-dumping, ε, πολιτική ανταγωνισμού, ε, κρατικές προμήθειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, βασικοί κανόνες για τις υπηρεσίες, ΦΠΑ και κανόνες για την ενέργεια που να σε ό,τι αφορά το εμπόριο της ενέργειας δηλαδή. Με αυτά το Ηνωμένο Βασίλειο εύκολα μπορεί να συμφωνήσει, μπορεί να συμμορφωθεί. Εκτός από αυτούς ε, που θέλουν ε, την απόλυτη έξοδο μέλη του UKIP δηλαδή κτλ. Σημαίνει Τώρα, τι σημαίνουν αυτά. Ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τι τελωνιακέ διαδικασίε και τα τεχνικά πρότυπα, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει στο πακέτο DCFTA ενδεχομένω να προσθέσουμε και την Τελωνιακή Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Ε, υπό την οικονομική συνεργασία. Ε, έχουμε διάφορα κεφάλαια που συνδέονται με το εμπόριο και κάποια που δεν συνδέονται με το εμπόριο. Αυτά που συνδέονται με το εμπόριο, ε, χρηματαγορέ, ε, ενεργειακή πολιτική, μεταφορέ, ε, κλίμα, προστασία των καταναλωτών ε, κοινωνικές πολιτικές και απασχόληση. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που η υπόθεση της Ουκρανίας περιλαμβάνει προϋποθέσεις για να δοθούν ε, κάποια διαβατήρια, ας πούμε, σε πολιτικές ε, που θα είναι αντίστοιχες με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Το κλίμα. Φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να συμμορφώνεται, να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις του Παρισιού, αλλά εδώ θα πρέπει να αποδεσμεύσει το ευρωπαϊκό κομμάτι της συμφωνίας ή να αποφασίσει να είναι τμήμα του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, ο Υπουργό Brexit πρόσφατα είπε ότι ε, μια και η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόληση δεν εμπόδισε το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει την πιο ευέλικτη αγορά εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βλέπει για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να κρατήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το βοηθάει για να αποφύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Υπάρχει και κάτι ακόμα σε αυτό το στην οικογένεια κεφαλαίων που είναι πολύ σημαντικό για το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι για το εμπόριο, αλλά αφορά επιστημονική έρευνα για την ενότητα εκπαίδευση το ορίζοντα 2020, το τέμπους και τις πολλές υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξαιρετική σημασία όλα αυτά. Η Συμφωνία Σύνδεσης παρέχει μια εγγύηση διαβεβαίωση ότι όλα αυτά θα ε, διαπραγματευθούν, θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευση. Υπάρχουν και άλλα τρία σημεία που δεν στη Συμφωνία Σύνδεση που είναι δύσκολα και που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Το πρώτο είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα θέλει να μην δεσμευτεί σε αυτό το τομέα. Και αν η Ευρώπη από την πλευρά τη πει ότι οι τέσσερι ελευθερίε πάνε πακέτο. Αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι θα πρέπει να δούμε αν η αρνητική έκβαση του διαλόγου για τον Brexit οδηγήσει σε επιστροφή πολλών μεταναστών και ενδεχόμενων μεταναστών που θα αποφασίσουν να μην πάνε τελικά στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε την αυθόρμητη μετανάστευση να πηγαίνει αντίστροφα, να έχει αντίστροφη ροή. Σε αυτή την περίπτωση η λίστα είναι πολύ απλή και συγκεκριμένα να αντιγράψουμε την ρήτρα διασφάλισης του 1999 της ε, Ελβετίας. ώστε να γίνει κάτι, χωρίς να να πούμε περισσότερα. Ε, βλέπουμε και άλλες πιο δύσκολες ε, δυνατότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ενδεχόμενη εξέλιξη, τώρα όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί εκπρόσωποι λένε ότι θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να πληρώσει. Δεν είναι σαφές ότι θα πρέπει να πληρώσει το Ηνωμένο για την ενιαία αγορά, για το ελεύθερο εμπόριο, για το DCFTA. Αυτό δεν είναι επίσης ξεκάθαρο. Το τελευταίο στοιχείο στον κατάλογο αυτό αφορά την ε, συνεργασία. Ακραίοι ε, υποστηρικτές ε, του Brexit ε, θέλουν να έχουμε ε, να έχουν αυτή την ε, απομόνωση στην να φτιάξουν νησί με 25% εταιρικό φόρο. Αυτό που αναμένω όμως είναι το Ηνωμένο Βασιλείο να πει ότι ενώ η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του 20% Πώς θα τεθεί αυτός ο όρος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεν θα μπορεί φυσικά γιατί είναι διαφορετικό το περιεχόμενο. Τα δύο άλλα χαρακτηριστικά της Συμφωνίας Σύνδεσης είναι κατά πρώτον είναι τα τεχνικά θέματα μιας συμφωνίας 2.000 σελίδων Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μειώσουμε τον χρόνο για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού και δεύτερο η ε, προσωρινή ρήτρα εφαρμογής με τη διατάξη του DCFTA που θα πρέπει να αποτελέσουν μια μεταβατική συμφωνία. Το θέμα αυτής της μεταβατικής συμφωνίας έχει θυχτεί από, τον, ε, από την Πρωθυπουργό δεν μπορώ να φανταστώ ποιο θα είναι όμως το νομικό περιεχόμενο. Με προβληματίζει αυτό και πέρα από τα σημεία που ανέφερα για την προσωρινή εφαρμογή και την ενδεχόμενη παράταση ε, στα δύο χρόνια για την θέση του άρθρου 50. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο μοντέλο που έχει δυναμική Είναι ένας κατάλογος που πρέπει να δούμε και θεωρώ ότι είναι η πιο κατάλληλη αναφορά αυτό το μοντέλο σύνδεσης από άλλα πιο παλιά, παλαιότερα και πιο γνωστά μοντέλα. Ευχαριστώ πολύ. I just Θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχουν άλλες δύο πτυχές στη Συμφωνία της Ουκρανίας που είναι πολύ χρήσιμες. Πρώτον, Υπάρχει ένας θεσμικός μηχανισμός ο οποίος περιλαμβάνει ετήσιες διασκέψεις, υπουργικά συμβούλια, τεχνικές επιτροπές, για τις οποίες έκανε λόγο και ο Μάικλ, κοινέ κοινοβουλευτικές επιτροπές, και ο δεύτερος όρος είναι ότι υπάρχουν ρήτρε για πολιτική συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Και για την εσωτερική ασφάλεια. για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανισμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται Στην Ουκρανία αυτό δημιούργησε πρόβλημα. Στην Ολλανδία υπήρξε πρόβλημα σε σχέση με αυτό και έγινε δημοψήφισμα για τη συγκεκριμένη πολιτική ρήτρα. Όμως προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα προκύψει πρόβλημα Θεωρώ ότι είναι ένας μηχανισμός για να συνεχίσουμε την εξαιρετική πολιτική συνεργασία που πετύχαμε μέχρι στιγμής. Τα τελευταία 40 χρόνια συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο Σέφλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Δύο σκέψεις δύο ερωτηματικά που μπορείτε να προσθέσετε στο τέλος. Όπως το βλέπω, το Ενωμένο Βασίλειο εμπλέκεται σε μία κρίση, σε δύο κρίσεις. Η σχέση του Ενωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και το άλλο είναι τι είδους Ενωμένο Βασίλειο θα προκύψει από αυτό. Βλέπω μια συνταγματική κρίση. Είναι ξεκάθαρο. Έχει να κάνει με την Βορειολανδία με το Γιβλα... και το Γιβραλτάρ. Δεν μπορώ πώς μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ούτως ή άλλως θα στερέψετε από πετρέλαιο, οπότε δεν έχει σημασία. Αλλά από ό,τι βλέπω ότι από την Σκοτία υπάρχει μια πιο αυστηρή γραμμή από την Νικόλα Στέρτζον. θα υπάρξει αντίθεση με τις, ε, αντίφαση με τις ε, συνθήκες και αυτό θα δημιουργήσει και θέματα ασφάλειας για τον Ηνωμένο Βασίλειο. Η ερώτηση μου είναι πότε θα ξυπνήσουν. Υπάρχει μια εφορία από όσο βλέπω. Θα ακολουθήσει και ένα hangover μετά από αυτήν την εφορία, είμαι σίγουρος. Πότε θα φτάσει η στιγμή που θα ξυπνήσουν και θα καταλάβουν τι έχουν κάνει. Θα υπάρξουν κραυγές προσδοσίας. Φαντάζομαι στην Daily Mirror τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πρόδωσε και πάλι». Μπρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους για τη συνεισφορά τους, η οποία ήταν πραγματικά ανεκτήμητη. Μας βοήθησαν να ρίξουμε φως και να διευκρινίσουμε πολλά ζητήματα. Αν κατάλαβα καλά για να συνοψίσω τις δύο σας προτάσεις. Να πω ότι καλώς πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνθήκη εξόδου μαζί με ρήτρα διασφάλισης άρθρο 50 και ενδεχομένως ήταν πρότασή σας πολιτικό κείμενο για το μέλλον της Ευρώπης που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε κείμενο Συμβουλίου για να μην είναι μεικτή συνθήκη πολιτική και θα πρέπει να ε, δουλευτεί αυτό το κείμενο με το Κοινοβούλιο παρόλο που θα εξεταστεί από το Συμβούλιο. Και στη συνέχεια να εξεταστεί ένα μοντέλο σύνδεσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα το πούμε ακριβώς. Όμως, ε, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε κύρωση ή επικύρωση από πλευράς κρατών μελών. Άρα, η προθεσμία θα ήταν πιο μεγάλη και γι' αυτό χρειαζόμαστε ρήτρα διασφάλισης για να καλύψουμε αυτή την περίοδο. Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω και ερωτήσεις. Πρώτον, το μοντέλο που είναι της Ουκρανίας, το προτιμάτε και δεν προτιμάτε μια συμφωνία τύπου Ελβετίας ή Νορβηγίας γιατί μιλούμε για χώρες πλούσιες και δυνατές, όχι μια χώρα που βοηθούμε όπως η Ουκρανία. Αν έχουμε θέσει αυτό το ερώτημα στην Ελβετία και στην Νορβηγία, δεν γίνεται να μην το θέσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, τα κρυφά επανεισάγουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις για την κατάσταση των εργαζομένων. Ό,τι βγήκε από την πόρτα το ξαναβάζουμε κρυφά από το παράθυρο. Σε κάθε περίπτωση θα τεθεί το πρόβλημα. Και πρέπει να τεθεί και το θέμα τι θα γίνει με την Σκοτία και την Ιρλανδία. Το πρώτο είναι πολιτικό, το δεύτερο θεσμικό. Γιατί οι Ιρλανδοί συνάδελφοι έχουν υπεθυμίσει ότι στη συνθήκη υπάρχει μια ρήτρα που δεν επιτρέπει την τροποποίηση εκτός εάν υπάρχει κοινή συμφωνία. Και η Ιρλανδία δεν θέλει να την τροποποιήσει. Άρα υπάρχει πολιτικό θέμα βούλησης γιατί ένα μέλος του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Λίγο κάπως διαφορετικά είναι τα ερωτήματα, δεν είναι ακριβώς ίδια. Σε κάθε περίπτωση, είτε μιλούμε για δημοψήφισμα, είτε για κάποιο άλλο μέσο επικύρωσης της συμφωνίας, θα πρέπει να διευκρινιστεί. Έχετε εκτίμηση, έχετε ε, κάποια άποψη για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Sorry, Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ πολύ, επόμενη ομιλήτρια. Είπα David, διακόπτη πρόεδρος, δεν είστε εσείς, δεν έχετε το λόγο, ο David έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σειρά μου δεν είναι. Καλώς, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Νταφ και κύριε Έμερσον για τις πολύ ενδιαφέρουσες σας παρουσιάσεις. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ακούγοντας διάφορους πολιτικούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, τι μαθαίνω. Μαθαίνω ότι λένε ότι θέλουν το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά, έχοντας φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοούν όταν, λένε, όταν μιλούν για πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά, ότι θα είναι μέλος της ε, ενιαίας αγοράς όπως η Νορβηγία. Ποιες άλλες δυνατότητες πλήρους προσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά υπάρχουν. Έχετε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό από ότι εμείς. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο. Ποια είναι η γνώμη σας για το εξή ενδεχόμενο. Μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η Βόρεια Ιρλανδία, όπως η Σκοτία, όπως το Γιβραλτάρ, να είναι μέλη του ΕΦΤΑ, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ή ακόμα και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Είναι αυτό εφικτό. Μιλούσα πριν από δύο εβδομάδες στο Λονδίνο με ένα σκοτσέζο πολιτικό υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτία. ήταν εκείνος και μου έλεγε ότι θα μπορούσε να συνδεθεί η Σκωτία 100% ή ακόμα και να μπει στην Ευρωπαϊκή ε, ε, Συμφωνία για το Ελεύθερο Εμπόριο, ακόμα και αν δεν είναι κυρίαρχο κράτος και ανήκει στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια είναι η θέση σα γι' αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώ Λάινεν. Σας ευχαριστώ πολύ για τις καινοτόμες προτάσεις. Ο Κίφερ Χόφστατ είναι ο βασικός διαπραγματευτής και μπορεί ίσως καλύτερα να ε, αντικατοπτρίσει αυτές ε, τις ιδέες και να μιλήσει καλύτερα. Εάν δεν υπάρχει επίσημη έκθεση, παρόλα αυτά έχουμε το Think Tank που αναφέρει ότι από τις τέσσερις ελευθερίες οι τρεις είναι οικονομικές και η τέταρτη πολιτική και θα πρέπει να διαιρεθούν ή μπορούν να διαιρεθούν. Όμως γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί αυτή την υποχώρηση, να υποχωρήσει δηλαδή και να δεχθεί ότι αυτές οι τέσσερις ελευθερίες δεν αποτελούν ένα σύνολο, αλλά μπορούν να ε, διαιρεθούν ή να, ε, να ασχοληθούμε με αυτές κατά τμήματα. Ξέρετε, έχουμε βρει κάποια σημεία που θα μπορούσαν να συζητηθούν χωρίς όμως να υπάρχει διάκριση σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν θα έπρεπε να συγκρίνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ουκρανία. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα ζητήματα. Εάν δει κανείς την ισορροπία δυνάμεων, την οικονομική ισχύ, το καθεστώς των δύο χωρών βλέπει ότι δεν έχουν καμία σχέση. Υπάρχει και αιτήσια συνεδρίαση του Κοινοβούλου με το, με το Westminster. Ίσως ε, τελικά χρειαστεί βοήθεια το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πρόεδρος. Η κυρία Τζέιμς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που πήρα το λόγο προηγουμένως ενώ δεν τον είχα. Θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι σε συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και είναι σαν να έχουμε καινούριο κοσκινάκι μου αν θέλετε, γιατί η Επιτροπή αυτή ακούει αυτά που θέλει να ακούσει. Ότι είναι κατά νέα σχήματα μαντάτα για τη Βρετανία, αν φύγει από την Ένωση, οι διάφορες οργανώσεις στέλνουν τους εκπροσώπους τους να πάρουν το λόγο, να απευθύνουν το λόγο στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Οι συγκεκριμένοι δύο που έχετε φέρει ε, έχουν ειδικά συμφέροντα και είναι σαφέστατα ταγμένοι υπέρ της μίας άποψης. Χαίρομαι για αυτά που είπατε, τα είπατε πολύ ωραία και τα γράψατε πάρα πολύ ωραία. Ε, ε στρέφομαι στους δύο μιλητές, αλλά είναι μονομερής η οργάνωση αυτής της συνεδρίασης. Εάν δεν αναφέρετε και κάποιον που να λέει την άλλη άποψη, τότε κινδυνεύετε να πέφτετε συνέχεια στην παγίδα του να καταλαβαίνετε και να πιστεύετε μία και μόνη νοοτροπία. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του δημοψηφίσματος και αναγνωρίζετε όλοι φαντάζομαι ότι εγώ είμαι στρία, ε, έχω παραστεί σε περισσότερες από 60 εκδηλώσεις και γεγονότα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, και μίλησα κατά. Άλλοι μιλούσαν υπέρ. Σε κάθε περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και όσοι ήμασταν υπέρ και όσοι ήμασταν κατά, είχαμε τον ίδιο χρόνο να, να μιλήσουμε στη διάθεσή μα. Οι συναντήσει ήταν αμερόληπτε, γιατί και οι δύο απόψει εκπροσωπούνται επαρκώ και με αντικειμενικό τρόπο και με δικαιοσύνη. Ε, αυτό δεν ισχύει εδώ πέρα στη σημερινή συνεδρίαση και δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσει να γίνεται κάτι τέτοιο. Να καλείτε δηλαδή ανθρώπους που παρουσιάζουν μόνο μία πλευρά ε, των πραγμάτων. Ε, ζητήθηκε ένα φιλικό διαζύγιο. Εμείς θελήσαμε να απεμπλακούμε από τον πολιτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε φορά που έχω παραστεί σε τέτοιου είδους παρουσιάσεις το, τα μόνα πράγματα που ακούω είναι εκδίκηση, κατηγορία εναντί του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή ήταν κακό παιδί, τιμωρία του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή ήταν κακό το Ηνωμένο Βασίλειο, αρνητικό και όχι προς τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέτοιου είδου ε, φρασιολογία χρησιμοποιείται. Ας ακούσουμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση παρακαλώ. Σα προειδοποιώ τα διεθνή μέσα επικοινωνίας και τα μέσα επικοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου ε, αναπαράγουν αυτές τις απειλές και αυτές δεν είναι προ όφελο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εκπλήσεστε που υπερασπίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας λέω ότι τα αναπαράγουν αυτά τα διεθνή μέσα Επικοινωνίας, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ισορροπημένη προσέγγιση του θέματος. Οι συνάδελφοι από το Sinn Féin κατέληξαν σε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για τα σύνορα στη Βόρειο Ιρλανδία. Είναι μια ποιοτική συζήτηση, ένας ποιοτικός διάλογος αυτός και θα ήθελα κάτι τέτοιο να γίνει και εδώ στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Μίλησε και ο κύριος Λάινεν για αυτά. Είναι καλό να έχουμε μια καλή οπτική γωνία, επαρκή εκπροσώπηση του ε, ε, του στρατοπέδου που είναι υπέρ της αποχώρησης και επαρκή εκπροσώπηση του στρατοπέδου που είναι υπέρ της παραμονής. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ θετική ανατροφοδότηση να σας δώσω. Και γι' αυτό λέω, ας σταματήσουμε αυτό το μονόλογο που τον έχουμε κάνει καραμέλα της καταδίκης του Ηνωμένου Βασιλείου και της εκδίκησης αυτού για την απόφαση που τόλμησε να πάρει. Θα σας ενημερώσω, επειδή πρόσφατα άρχισατε να έρχεστε στις συνεδριάσεις μας, να σας πω ότι στις συνεδρίες των συντονιστών το συζητήσαμε διαμακρών το θέμα και συμφωνήσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, όχι μόνο τώρα, τους επόμενους μήνες και χρόνια ανάλογα με το πόσο γρήγορη ή αργή θα είναι η διαδικασία Brexit. Και όλοι οι συντονιστές θα μας δώσουν ονόματα εμπειρογνωμόνων που θέλουν να έρθουν εδώ για να μιλήσουν σε αυτές τις ε, συζητήσεις. Η πολιτική σας ομάδα δεν μας έδωσε κανένα όνομα. Ακούσαμε λοιπόν ε, τους ε, εμπειρογνώμονες που πρότειναν άλλοι συντονιστές. Αλλά σας καλούμε και η δική σας πολιτική ομάδα να προτείνει ε, κάποιον εμπειρογνώμονα, η Μαρτίνα Άντρεσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από αυτά που είπε ο Τζόρτζ, θα ήθελα να πω κάτι κι εγώ για πιθανή συνταγματική κρίση στα πλαίσια της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Είναι σημαντικό η Επιτροπή σας και οι εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με αυτό το θέμα να καταλάβουν ότι η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, που ήταν μία συμφωνία που οδήγησε στα δύο δημοψηφίσματα στην Ιρλανδία, Μόρια Ιρλανδία και Νότια Ιρλανδία, δηλώνει ότι όλοι οι θεσμοί και οι συνταγματικές διευθετήσεις, ε, η συνέλευση κτλ., ε, όλοι οι φορείς της Ιρλανδίας και οποιασδήποτε τροπολογίες στην Βρετανική πράξη το Σύνταγμα της Ιρλανδίας, όλα αυτά με το Σύνταγμα της Ιρλανδίας είναι αλληλένδετα. Μια και οι δύο κυβερνήσεις είναι συνεγγυητές της συμφωνίας της, συμφωνίας της ε, Μεγάλης Παρασκευής, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Θα πρέπει να δούμε το ειδικό καθεστώς της Βόρειας ε, Ιρλανδίας, ούτως ώστε να μπορέσει να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά κανένα κρατός μέλος δεν έχει φύγει ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Και θα πρέπει να, δούμε, να βρούμε ενδεχομένως εφάνταστες λύσεις. Αυτό που θέλω να κάνω έκκληση όμως στο Ευρωκοινοβούλιο είναι να μην στρέψει την πλάτη στον Ιρλανδικό λαό, ο οποίος έχει περάσει μια φοβερή σύγκρουση και εγώ ήμουνα τμήμα αυτής της σύγκρουσης, πληγώσαμε ένα τον άλλον, έγινε μια τεράστια προσπάθεια συμφιλίωσης, η οποία συνεχίζεται και δεν θέλουμε να δούμε μια γενιά νέων ανθρώπων οι οποίοι μας κοιτάνε αυτή τη στιγμή, έχουν το βλέμμα στραμμένο πάνω τους, με ένα ψήγμα έτσι κατηγορίας. Εσείς μπορέσατε, είχατε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι. Και τώρα αυτό που αντιμετωπίζουμε, το φάσμα που αντιμετωπίζουμε είναι την ενίσχυση του διαχωρισμού. Σκεφτείτε την καταστροφή που θα κάνει αυτό στην Ιρλανδία και στην ειρηνευτική διαδικασία. Σήμερα κοίταξα κάτι που είπε ο πρόεδρος Μπαρόσο, γιατί έχει δημιουργήσει την ε, Task Force Μπαρόσο όταν ήταν επίτροπος. Και είπε ότι η ειρήνη στην ε, Ιρλανδία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί στην Ευρώπη υπάρχει μάλλον η ευρωπαϊκή διάσταση, μια και οι πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Όλοι έχουμε Ιρλανδικά διαβατήρια, άρα είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένων των τριπτικών αρχών της ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, που είναι η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ειδικά προβλήματα ε, Βόρειας Ιρλανδίας, Σκοτίας, που ψήφισαν κατά συντριπτική πλειοψηφία να παραμείνουν. Και Γιβραλτάρ το ίδιο. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου ένα τμήμα της Ιρλανδίας είναι εντός και ένα τμήμα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μην ξεχνάτε, θα έχετε δυσκολίε και με την αγορά. Πώ θα σταματήσετε, α πούμε, του λαθρέμπορου. Πώ θα σταματήσετε έξι κομιτείε ε, όταν έχουμε ε, σύνορα 350 μίλια. Αν παραδείγματο χάρη η Βρετανία φύγει και ε, τελικά η Βρετανία έχει μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία, με, με, με, με διάφορες χώρες, ό,τι και να εξασφαλίσουν οι εμπορικές συμφωνίες, δεν θα έχουν τα ίδια ρυθμιστικά, τις ίδιες ρυθμιστικές επιπτώσεις με αυτό που έχουμε εμείς. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί, θα περιφέρονται στα σύνορα, θα μπαίνουν στην ενιαία αγορά και εν συνεχεία από κράτος σε κράτος θα, θα πηγαίνουν από το ένα κράτος στο άλλο, μια και δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα κοινή περιοχή για τους ταξιδιώτες θα πρέπει να προστατευτεί. Εγώ μίλησα ευρωβουλευτές που, με ευρωβουλευτές που είπαν ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ενιαία αγορά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ας πούμε, στους λαθρέμπονους αυτοκινήτων να κάνουν ανενόχλητη τη δουλειά τους. Πρέπει να καταλάβουμε τις επιπτώσεις ε, ενός διαχωρισμού. Επομένως, χρειάζεται ε, ένα ειδικό καθεστώς Δεν μπορείτε να προτείνετε κάτι και να πείτε «Να, αυτό είναι, δούλεψε εκεί, να το χρησιμοποιήσουμε». Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ κάποιο κράτος μέλος δεν έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τους μηχανισμούς. Να βάλουμε δηλαδή, να σκεφτούμε και να βρούμε φάνταστες λύσεις ε, για να δούμε πώς θα γίνει ε, και πώς θα ρυθμίσουμε το πρόβλημα της Ιρλανδίας. Λοιπόν, ο Μάικλ Έμερσον και ο Άντρου Νταφ να απαντήσουν μετά από τις ε, ερωτήσεις που ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας στον Τζόρτζ Σεφλίν για τη Σκότια και την κυρία Άντερσον. Είμαι Άγγλος με σκοτσέζικο αίμα και βορειοελλανδικό αίμα στις φλέβες μου, οπότε είναι επόμενο το αυτό και για εμένα. Όσον αφορά αυτό που ο Τζόρτζ για τη Σκωτία, δείξαμε αυτοσυγκράτηση στο θέμα της σχέσης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ενωμένο Βασίλειο. Το θέμα της Βόρειας Ιρλανδίας είναι διαφορετικό γιατί υπάρχει πρόβλημα στα σύνορα και επειδή είναι πολύ σχετική και η πρόταση για την Τελωνική Ένωση και επίσης θα έπρεπε να αναφέρω και την υποθετική συμφωνία σύνδεσης θα έχει και ένα στατικό για την ε, ελεύθερη κυκλοφορία πρώην Υπουργό Εσωτερικών την προηγούμενη, ε, την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι τα 32 σημεία στα οποία όπτην τον προηγούμενο χρόνο του Ηνωμένο Βασίλειο θα τα συνεχίσει. Αυτά αφορούν την, τα θέματα ασφαλεία αυτά τα 32 σημεία. Τον κύριο Ρούσο, όσον αφορά την επικύρωση και την, ε, στην κυρία Μπρεσό μάλλον, η καθυστέρηση ε, η ενδεχομένη μπορεί να είναι δύσκολη. Η προσωρινή εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε χωρίς να περιμένουμε την επικύρωση. Το σχόλιο που κάνετε για το μοντέλο που προτείναμε και το κατά πόσο ανταποκρίνεται σε αυτό της Νορβηγίας και της Ελβετίας είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Για μένα είναι ανοιχτό το ερώτημα. Ως προς το κατά πόσο αυτό αποκρίνεται θα μπορούσε να πει κανείς ότι η συμφωνία σύνδεση και το περιεχόμενό της, αν δούμε τον κατάλογο του κεκτημένου, βρεβού κεκτημένου που περιλαμβάνεται, όπως δεν ε, είναι σαν το... E e σαν της ΕΟΧ, δεν υπάρχει τόση επιλεκτικότητα Παρέρχομαι στο θέμα της Σκοτίας και στη μετανάστευση. Ο Πρωθυπουργός της Σκοτίας είπε ότι μπορεί να είναι μια αποκεντρωμένη, ε, να έχει ε, αποκεντρωμένη δικαιοδοσία η Σκοτία για τη μετανάστευση. Αν δει κάτι τέτοιο το Βασίλειο στην Σκοτία, μπορεί να μην, έχει, να μην συμφωνεί με κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείω την ιδέα αυτή για το θέμα της μετανάστευσης. Μπορούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει σχετικά με αυτό. Όσον αφορά την πλήρη πρόσβαση, η διατύπωση που χρησιμοποιείται ε, από την Πρωθυπουργό είναι η μέγιστη δυνατή πρόσβαση, όχι η μέγιστη πρόσβαση γιατί δεν τους αρέσει το μοντέλο της Νορβηγίας. Γιατί είναι πολύ κοντά στην πλήρη συμμετοχή. Θα μπορούσαν ενδεχομένω η Σκωτία και το Γιβραλτάρ να κάνουν μια συμφωνία 7, τύπου 7. Σε αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι όχι. Θα πρέπει να είναι κυρίαρχο κράτος κάποιο για να μπορέσει να ε, κάνει συμφωνία στο πλαίσιο της 7. Θα πρέπει να βρούμε μια πιο εφάνταστη λύση. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή, όμω αυτή είναι η πρώτη απάντηση που μπορώ να σα δώσω σε αυτό το ερώτημα. Για τι τέσσερι ελευθερίε. Δεν κάνω κάποια πρόταση από αυτού. Περιγράφω κάποια σενάρια για το πώ θα προχωρήσουν οι ε, διαπραγματεύσει. κυρία Τζέιμς που από ό,τι φαίνεται έχει φύγει, από ό,τι βλέπω έφυγε, Προσπάθησα να μην ε, εκφράσω προσωπική άποψη για τα θεμελιώδη ε, θέματα. Προσπάθησα να είμαι ένα πειθαρχημένο ερευνητή. Όμω αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι καμία συμφωνία, εμπορική συμφωνία στον κόσμο, εκτό από τη συμφωνία ΕΟΧ με την Νορβηγία, δεν περιέχουν όρο για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Υπάρχουν πάρα πολλές συμφωνίες με πολλές τρίτες χώρες, δεν περιλαμβάνουν τέτοιου είδους όρος. Είναι ειδική περίπτωση βέβαια του Ηνωμένου Βασιλείου, πράγματι. Αλλά ε, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, όπως βλέπετε, που θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε ε, να βρούμε ε, μια διέξοδο αν υπάρξει αυτόματη ε, ε, μείωση της μετανάστευσης. Τότε το μοντέλο του 1999 της Ελβετίας που είναι σύμφωνα με, το με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα μπορούσε να δώσει τη λύση στο πρόβλημα, να τραγωνίσει τον κύκλο. Ευχαριστώ. Um, uh, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα, μάλλον με συγχωρείτε. Πρώτα, θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στην κυρία Τζέμις που δεν είναι παρούσα αυτή τη στιγμή. Είπα ότι έχουμε προσωπικό συμφέρον σε αυτό το θέμα. Είμαι παρτιζάνο και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν εδώ. Αλλά δεν είναι ευγενικό εκ μέρου τη και ειδικά το γεγονό ότι έφυγε πρωτού προλάβω να δώσω την απάντηση. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω με έναν πυρογνώμονα από το UKIP. Πραγματικά θα ήθελα να μπορέσω να, δια... να μιλήσω με κάποιον που θα ξέρει γιατί πράγμα μιλάει και που θα ανήκει στο αντίπαλο στρατόπεδο. Αν μπορέσετε να τον οργανώσετε, ευχαρίστω να είμαι και πάλι παρόν. Τώρα, όσον αφορά τη Σκοτία, η Νίκολα Στέρτζεν είπε ότι θα συμφωνήσει με την ε, απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι θέλει να συμπεριληφθεί επειδή υπάρχει αυτή η διαφωνία με το Λονδίνο, με την κεντρική κυβέρνηση. Και όσον αφορά το ευρύτερο ερώτημα, το αντικτύπου του Brexit στην ε, σύνθεση σύνθεση του Ηνωμένου Βασιλείου και των ε, Βρετανικών νήσων, θεωρώ ότι δούμε σε μια ευρύτερη ε, ομοσπονδιακή δομή εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και θα υπάρξει περαιτέρω αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων από το Λονδίνο. Όμως η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε ότι το Ενωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση. Συμφωνάμε με αυτά που είπε ο Μάικλ. με την ε, ποικιλομορφία που υπάρχει στα διάφορα καθεστώτα σύνδεσης. για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων. Φυσικά και θα υπάρχει, αλλά θα είναι στην ίδια βάση που σημαίνει αυτό και με την Ουκρανία. Είναι σαφές από τις δηλώσεις της Πρωθυπουργού ότι για να κάνει το κόμμα της να αποδεχτεί για να προοπτική για τον Ηνωμένο Βασιλείο δεν θα πρέπει να αποκλείσει αυτό. Στη συνθήκη υπάρχει το άρθρο 8 το οποίο κάνει λόγο για στενή εταιρική σχέση με προβληματικούς γείτονες. Έχει συμπεριληφθεί αυτό στο συνθήκη της Λισαβόνας επειδή ακριβώς η Ήπειρος γινόταν όλο και πιο περίπλοκη, η μορφολογία ήταν πιο περίπλοκη σε σχέση με το παρελθόν. θα πρέπει να μείνουμε πιστοί στην συνθήκες Λισαβόνας αναφορικά με αυτό. Να μην δημιουργήσουμε τριβή. Πρέπει να πετύχουμε το αντίθετο από αυτό. Έχουμε προβλήματα, ναι, αλλά με σκληρή δουλειά και με θετική πολιτική βούληση νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μία συμφωνία που θα είναι σεβαστή και από τις δύο πλευρές και που θα είναι μόνιμη. Κάνατε μία ερώτηση για το ποιος είναι ο αρμόδιος, ποιος είναι εκπρόσωπος για αυτά τα θέματα ε, στην κεντρική κυβέρνηση. Η ειλικρινή ερώτηση, απάντηση στην ερώτηση είναι ότι απλώς δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά από τη μία πλευρά και από την άλλη να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε. Πρέπει ο κ. Φερχόφστατ να πάει και να το κάνει αυτό. Αυτό θα πρέπει να πάει και να του εκπαιδεύσει. και στη Βουλή των Κοινωνιτών υπάρχει μια ειδική επιτροπή για τον Brexit. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, αλλά θα ήταν κάτι που έπρεπε ενδεχομένω να το δοκιμάσουμε και στη Βουλή των Λόρδων. Υπάρχει μια... Ε, υπάρχουν 30 ερωτήματα στη Βουλή των Λόρδων που έχουν να κάνουν με τις διάφορες πτυχές αυτού του προβλήματος που έκυψε με το Brexit. Πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση στο θέμα, κατά την άποψή μου. Και θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, σε αυτό το θέμα. είναι η αρχή μιας μακράς διαδικασίας. Θα υπάρξουν επιπλογές, έντονες διαφωνίες, αλλά το πρότυπο αυτό, το φορμάτ που περιγράψαμε και παρουσιάσαμε είναι κάτι έξυπνο. Θα πρέπει να το ε, συλλογιστούμε. Θα θέλετε να πείτε κάτι και ε, κάτι για τα, τις επενδύσεις, τα προσωπικά συμφέροντα που έχετε. Ναι, απαντώ λέγοντας ότι εισπράττω σύνταξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πρώην βουλευτής. Και ναι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προσωπικό συμφέρον. Ευχαριστώ. Άρα στις διαπραγματεύσεις συμφωνείτε ότι θα πρέπει να αμυφθείτε από το Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και αν υπάρξουν καινούργιες σκέψεις θα μας τροφοδοτήσετε με αυτές. Είστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι και οι δυο σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Θα τα πούμε στις 21 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο στις 7 και στις 29 Νοεμβρίου πλήρης ημέρα συνεδρίασης.